Καλημέρα σας. Euh, καλημέρα σας. Ε, έχουμε μια ανακοίνωση από πλευρά των διερμηνέων. Ε, σας, ε, οι διερμηνείς σας, σας πληροφορούν με τα λύπης ότι συνεχίζει η εργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι νέε συνθήκε εργασία, πράγμα που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίηση για απεργιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα τη ερμηνεία για του Ευρωβουλευτέ και του Ευρωπαίου πολίτε κινδυνεύει. Δυστυχώ, λόγω τη εργασιακή διαμάχη, η διερμηνία θα σταματήσει ακριβώ στι 12.30 όπω προβλέπει το πρόγραμμα τη συνεδρίαση. Και τώρα το διαδικαστικό του κυρίου Λούντγκρεν. Ε, τη Δευτέρα βάλατε τη συζήτηση για το δικό μου θέμα που δεν θα μπορέσω να είμαι εδώ. Αυτό διακυβεύει την πολιτική μου αξιοπιστία. Σας παρακαλώ πολύ μην βάζετε ψηφοφορία τη Δευτέρα γιατί είναι μέρα μετακίνησης για όλους τους ευρωβουλευτές και έχουμε πάρα πολλά προβλήματα με ακυρωμένες και καθυστερημένες πτήσει. και είναι πολύ δύσκολο να φτάσουμε εδώ. Παρακαλώ λοιπόν στο μέλλον να το λαμβάνετε αυτό υπόψη, να μην βάζετε τις ψηφοφορίες σε μια ημέρα ταξιδιού. Ε, πρόεδρος, συμφωνώ. Κατάλαβα τι θέλατε να πείτε, αλλά νομίζω πως ε, πρόκειτο... για Κάτι που συζητήσαμε και με τους συντονιστές, αλλά συμφωνώ, θα το ε, θίξω και εγώ ξανά, γιατί πρόκειται για σημαντική ψηφοφορία και να μην μπαίνουν αυτή τη Δευτέρα. Αναμένοντας λοιπόν, συμφωνώ αγαπητέ Πίτερ, όπως σας είπα, περιμένοντας την αγαπητή μας ε, Πρόεδρο θα πρέπει να αρκεστείτε στον ε, μιστακοφόρο ε, και γυρεότερο Πρόεδρο και για να ξεκινήσουμε τις εργασίες μας. Δεν είμαι τόσο ευχάριστος, αλλά τι να κάνουμε. Περάστε όπως περνάτε τώρα. Ε, τώρα Φαντάζομαι πως όλοι λάβατε κάποιο email από πλευρά των διερμηνέων. Πρόκειται για την ανακοίνωση που σας ε, διαβάσαμε. Γίνεται κάποια διαπραγμάτευση ε, για ε, εργασιακά προβλήματα. Και οι διερμηνείς μας ζήτησαν να σας διαβάσουμε ένα σύντομο μήνυμα στην αρχή της συνεδρίασης. Και αυτό το σύντομο μήνυμα τετλοφορείται «Όχι υπέρβαση». Οι διερμηνεί σα πληροφορούν ότι συνεχίζεται η εργασιακή διαμάχη με τη διοίκηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τι νέε συνθήκε εργασία που αποτέλεσε το αντικείμενο προειδοποίηση για απεργιακή κινητοποίηση. Η ποιότητα τη διερμηνία ε, για του Ευρωβουλευτέ και του Ευρωπαίου πολίτε κινδυνεύει. Λόγω της εργασιακής διαμάχης, δυστυχώς η διερμηνία θα σταματήσει στις 12.30 ακριβώς, όπως προβλέπει το πρόγραμμα της συνεδρίασης και δεν θα υπάρξει καμία περίοδος χάριτος, δηλαδή προσθέτει ο Πρόεδρος. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να μείνουμε εντός του ωραρίου. Το βασικό ήταν να επιστήσουμε την προσοχή σας σε αυτήν την διαμάχη και την πιθανή υλοποίηση της απειλής για απεργία των διερμηνέων, πράγμα που θα διαταράξει τις εργασίες μας όπως καταλαβαίνετε. Να προχωρήσουμε τώρα στο σχέδιο της για τα ε, ε, και να σας ρωτήσω αν την εγκρίνετε. Έχουμε και τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 25ης Απριλίου και της 14ης και 15ης Μαΐου του 2018 που έχουν ε, συναυθεί στα in Εγκρίνονται αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Ανακοιώσει της Προέδρου δε, ή του ούτε του Αντιπροέδρου δεν υπάρχουν. κατά συνέπεια μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι οι λιμενικές εγκαταστάσεις ε, ε παραλαβής αποβλήτων του ε, πλοίων. Θα δώσω λοιπόν το λόγο καταρχάς στην Επιτροπή που θα μας παρουσιάσει το έγγραφο και μετά στην εισηγήτρια κυρία Μέισνερ στους κοιόδες εισηγητές και στη συνέχεια στους βουλευτές που θα θελήσουν να πάρουν το λόγο Έχετε λοιπόν το λόγο εξ ονόματος της Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλημέρα και στους διερμηνείς και σας ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την πρόταση αναθεώρησης και μια νέα οδηγία για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων. Σε δύο λεφτά θα έχετε και τις διαφάνειες. Και αν όχι θα ξεκινήσω να σας μιλάω και μετά θα θα δείτε και τις διαφάνειες. Νομίζω πως κάτι γίνεται με τις ε, διαφάνειες. Εν πάση περιπτώσει, όπω σας είπα, είναι ένα νέο κείμενο, αλλά στην ουσία πρόκειται για αναθεώρηση της οδηγίας, ε, της οδηγίας που καταθέσαμε από το 2000, ε, που όμως προτάθηκαν τόσες αλλαγές που θεωρήσαμε ότι θα ήταν ευκολότερο να φτιάξουμε τελείω νέο κείμενο. Ο στόχο δεν άλλαξε σε σχέση με τον αρχικό που ήταν ε, δηλαδή να μειωθεί ο φόρτος των αποβλήτων από τα πλοία και των ε, υπολείπων από τα φορτία ε, που ρίπτονταν στη θάλασσα. Αυτό σε συσχέτιση και με την συμφωνία Μαρπόλ για την πρόληψη της ρήπανση τη θάλασσα από τα πλοία. Προτείναμε λοιπόν να καλυφθούν όλα τα σκάφη και τα μικρά αλλιευτικά και τα σκάφη αναψυχή, καθώ και όλες τις εκθέσεις να συντάσσονται από τα ποντοπόρα πλοία. Ε, ε, έχουμε προσθέσει διάφορα στοιχεία που θεωρούμε πως ήταν πιο αποτελεσματικά για την εφαρμογή και την επιβολή και αυτή είναι η βασική διαφορά ανάμεσα στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και το νομικό πλαίσιο του Διεθνούς, Οργανισμού Ναυτιλίας ώστε η επιβολή να γίνεται στα πλοία σημαία και στο δικό μας πλαίσιο η εφαρμογή του, της νέας νομοθεσίας επί της οποίας συμφωνεί Κοινοβούλιο και Συμβούλιο. Αυτή η πρόταση εμπίπτει στο ευρύτερο πλαίσιο της περιβαλλοντικής και από άποψη χρονική σύμπτωση, ε, είδε το φω τη ημέρα ταυτόχρονα με τη δέσμη τη κυκλική οικονομία, αλλά και τη στρατηγική για το πλαστικό που προτείναμε κάποιου μήνε αργότερα που συνδέονται μεταξύ του. Ε, συνεργαστήκαμε με τι άλλε υπηρεσίε, ώστε να ε, διασφαλίσουμε ότι όλα εντάσσονται σε μια συνολική πολιτική που θα εξασφαλίσει καθαρότερο θαλάσσιο περιβάλλον και προστασία των θαλασσών γύρω από την Ευρώπη σε ολόκληρη την Ευρώπη. Διαφάνειες τώρα. Ξεκινήσαμε με μια εμπεριστατωμένη αξιολόγηση του νομοθετικού πλαισίου όπως είχε θεσπιστεί και γι' αυτό και ήταν αρκετά θετικό το ότι φτάσαμε σε μια πρόταση με ένα refit του 2015. Καταρχάς ήταν σαφές ότι χρειαζόταν αναθεώρηση της ισχύουσα οδηγία μέχρι τότε και εντοπίσαμε καταρχάς ότι η διαθεσιμότητα ε, λιμονικών εγκαταστάσεων παραλαβή στο θέμα της παράδοσης αποβλήτων σε αυτές τις εγκαταστάσεις και το διοικητικό φόρτο σε σχέση με την εφαρμογή και την επιβολή. Ο φόρτο βαραίνει τι δύο πλευρέ, δηλαδή τόσο το πλοίο όσο και του διοικητικού φορεί των λιμένων. Δεν θα σα κουράσω με τι λεπτομέρειε του εγγράφου, αλλά ίσω κάτι που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι μετά την τελική απόφαση να ευθυγραμμιστούμε όσο γίνεται περισσότερο με τη σύμβαση Μαρπόλ, με ιδιαίτερη εστίαση στα θαλάσσια απόβλητα, ήταν γιατί θεωρήσαμε πως οι αλλαγές στη Σύμβαση Μαρπόλ ακολουθούν το σωστή πορεία και εντάσσονται στο πλαίσιο της γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής όσον αφορά το θαλάσσιο περιβάλλον και τη λειτουργία των, της ναυτιλίας των θαλασσίων μεταφορών. Θέλαμε όμως να βελτιώσουμε ακόμη περισσότερο τη δική μας πρόταση. Όπως σας είπα, η πρόταση έχει μια, ένα διπλό στόχο. Ο εν, πρώτος είναι να περιοριστεί ο φόρτος αποβλήτων από τα πλοία και δεύτερον να διευκολυνθούν οι θαλάσσιες μεταφορές. Και πάντοτε θα πρέπει να εξετάζουμε την πρόταση αυτή έχοντας υπόψη αυτούς τους δύο κεντρικούς στόχους. Εάν δούμε και την κυκλική οικονομία, Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οτιδήποτε εμπίπτει στην κυκλική οικονομία θα αντικατοπτρίζεται κατά κάποιο τρόπο και στην πρόταση αυτή. Εδώ θα αναφέρω τη συμβολή των βεγών ε, ε, ε, αποβλήτων από τα πλοία στο γενικότερο πρόβλημα των αποβλήτων, τα σκάφη όλα που πρέπει να καλύπτονται από την οδηγία και έπειτα την, τον, τον ευάλωτο χαρακτήρα και το περιβάλλον διαφόρων θαλασσίων λεκανών. Αυτό είχε ενταχθεί αρχικά μέσα στη ε, μελέτη αντικτύπου την ε, περιφερειακή, γιατί είχαμε ήδη καταλάβει ότι έπρεπε διαφορετικά να δούμε τις διάφορες θαλάσσιες λεκάνες ε, της Ευρώπης. Αν δείτε τώρα τις διατάξεις της οδηγίας, καταρχάς έχουμε το θέμα της καταλληλότητας των εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων στους λιμένες, διευκόλυνση και αύξηση των οικονομικών κινήτρων και εξαιρέσεις. Να συγχωρείτε, λέει ο και τέλος έχουμε και κάποιες διοικητικές διατάξεις εντός της οδηγίας. Αν δείτε τώρα το θέμα της καταλληλότητας, ε, εξετάζουμε τον ορισμό που προτείνεται ε, με τις κατευθυντήριες γραμμές του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας ε, μένουμε κοντά στο διεθνή κανονισμό, διότι η οδηγία αυτή φυσικά θα ισχύσει για όλα τα σκάφη, άσχετα από τη σημαία που φέρουν, άσχετα από το λιμάνι προέλευση από τη στιγμή που πιάνουν σε ευρωπαϊκό λιμάνι. Επίσης περιλαμβάνεται μια νέα κατηγορία αποβλήτων που είναι τα κατάλοιπα από, την, ε, από τον καθαρισμό ε, και επίσης ε, περιλαμβάνεται, συμμορφωνόμαστε προς την απέτηση διαχωρισμού των αποβλήτων πάνω στο, λιμα, πάνω στο πλοίο ε, ε, γιατί αυτό συμμορφώνεται με τη γενικότερη οδηγία για τον διαχωρισμό των αποβλήτων και επίσης καλούμε για διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους χρήστες. Αυτό εν μέρη αντικατοπτρίζει αυτά που έχουμε βάλει και στο κανονισμό για τα λιμάνια, όπου καλούμε τα λιμάνια να διαβουλευθούν με τους χρήστες για τις διάφορε υπηρεσίες που προσφέρουν. Τώρα, όσον αφορά τα κίνητρα για την παράδοση και των αποβλήτων, η βασική αρχή είναι το δικό μας σύστημα ανάκτησης για αντιστοίχηση με το κόστος περιλαμβανόταν στο νέο Άνεξ 4 ε, επίσης έχει υπολογιστεί η σημαντική συνεισφορά που θα πρέπει αυτός ο υπολογισμός να ισχύει πάλι για όλα τα σκάφη. Ε, πάλι να επαναλάβω ότι η συμπερίληψη όλων των σκαφών είναι πολύ σημαντική εάν θέλουμε να πετύχουμε τους στόχους της οδηγίας. Προτείνουμε 100% ε, έμεσο τέλος για τα, για τα σκουπίδια που εκεί θα περιλαμβάνονται και τα παθητικά λιευμένα απόβλητα και οι ε, μηχανισμοί αλληλείας. Έχουμε εδώ όλα αυτά όπως σας είπα εντάσσονται στην πολιτική και το όραμα για τη ε, ε, μείωση και των πλαστικών αποβλήτων και όλα αυτά αναπτύσσονται με τον παρόμοιο τρόπο σε ολόκληρη την Ένωση. Προτείνουμε διαφοροποίηση για το τέλος ανάλογα με την κατηγορία, το είδος, το μέγεθος και το είδος της κυκλοφορίας του πλοίου ε, που πιάνει σε ευρωπαϊκό λιμάνι. Μετά για την επιβολή όσον αφορά το πεδίο της υποχρεωτικής παράδοσης. Έχουμε δεύτερη ευθυγραμμιστεί με τη Μαρπόλ. Έχουμε ε, ε παρόμοιες προσεγγίσεις. Εμείς, ε, η Μαρπόλ απαγορεύει την ρήψη των αποβλήτων. Εμείς βάζουμε την υποχρέωση παράδοσης στο λιμάνι. Είναι ακριβώς ο ίδιος στόχος, αλλά βλέπουμε ένα διαφορετικό τμήμα της επιχείρησης κάθε φορά. Γιατί με την υποχρέωση παράδοσης στα λιμάνια, στην ουσία ε, επιβάλλουμε αυστηρούς και προβλέψιμους μηχανισμούς επιβολής αυτής της οδηγίας. Προτείνουμε ε, να εξηγήσουμε και να υπολογίσουμε και να ορίσουμε πώς ε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί μία επαρκής ε, χωρητικότητα αποθήκευσης. Μιλάμε για αυτό το πράγμα μέσα στην οδηγία. Ε, μετά, πώς θα διευκολυνθούν οι αναφορές μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα λιμάνια. Οργανωμένη και συνολική συνολικό μάλλον καθεστώς για ελέγχους ε, στα σκάφη, στα λευτικά σκάφη ανάλογα με τα μεγέθη τους. Τώρα, εξετάζοντας τις εξαιρέσεις, έχουμε εξαιρέσεις σε σχέση με την, ε, ε, τα, με τα πλοία που κάνουν τακτικά δρομολόγια και πιάνουν τακτικά σε συγκεκριμένα λιμάνια, θεωρούμε πως ε, εδώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αναφοράς με πρακτικό τρόπο. Προτείνουμε εξαίρεση σε περίπτωση για ρύθμιση, ε, για παράδοση και πληρωμή σε κάποιο λιμάνι ε, με βάση την πορεία του πλοίου. Δηλαδή δεν χρειάζεται να παραδίδει απόβλητα σε κάθε λιμάνι, αλλά σε κάποιο από τα λιμάνια που θα πιάσει μέσα στην ευρωπαϊκή του ε, πορεία. Ε, ο στόχος είναι να αποφευθεί η ρήψη στη θάλασσα. Έχουμε ακόμα μια σημαντική αναφορά σε πιθανές αλλαγές της Μαρπόλ, στην περίπτωση της σύμβασης Μαρπόλ. Ε, αυτά εφαρμόζονται θα, εφαρ... θα ισχύσουν, αλλά έχουμε και μια ρήτρα ασφαλεία σε περίπτωση που αυτές οι αλλαγές, κάποιες από αυτές τι αλλαγές δεν συμφωνήσουν με τις... Ε, ε, ακριβώς με τις αλλαγές. Θα σταματήσω σε αυτά. Είμαι στη διάθεσή σας για να εξηγήσω τις προτάσεις και να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα την εισηγήτρια, αφού έχουμε ακούσει την Επιτροπή. Ζήνου. Η κυρία Μάισνερ, ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση της εκθέσεως. Όντως, όταν έρχονται προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, υπάρχει κάποια αναταραχή στο Κοινοβούλιο ή και στο Συμβούλιο όταν η ε, Επιτροπή προτείνει διάφορες τροποποίησεις. Φαίνεται ωστόσο ε, στην παρούσα πρόταση να περιλαμβάνονται πολλέ καλέ προτάσει ε, που βρίσκουν ευνοϊκή απήχηση και στι χώρε μέλη και στο Κοινοβούλιο. Άρα καλή αναθεώρηση. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ δεν θα κάνω και άλλε προτάσει αλλαγών. Καθαρά διαδικαστικά γνωρίζουμε ότι του χρόνου βεβαίω είναι οι ευρωεκλογέ και θα πρέπει να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία για διάφορου φακέλου μέχρι τότε. Ελπίζω θα είναι πάρα πολύ θετικό να μπορέσουμε να το προλάβουμε αυτό, διότι έχει μια γενική προσέγγιση έτοιμη το Συμβούλιο και νομίζω ότι και στο Κοινοβούλιο μπορούμε να φτάσουμε να ολοκληρώσουμε τη γνωμοδότηση μέχρι τέλος του φθινοπόρου, ώστε να προχωρήσουμε στους τριμερείς διαλόγους. Αυτό είναι και το σχέδιο, δηλαδή Αυστριακή Προεδρία, προώθηση και μετά Ρουμανική Προεδρία. Είχα πάει στην, στο λιμάνι της Κωνσταντσα και μου είπαν οι Ρουμάνοι, α, νομίζουμε ότι θα τελειώσει και στη δική σας Προεδρία, την Αυστριακή δηλαδή. Έχω βέβαια και επαφές με τους και οδησίγητες, αλλά ω τώρα δεν έχουμε συναντηθεί. Ήθελα σήμερα να κάνουμε μια συνάντηση, αλλά δυστυχώς ήμουν εκτός μάχης λόγω προβλημάτων μέσης, δηλαδή η, πονά, η μέση μου. Και θα δούμε, αλλά γνωρίζω καλά όλες και όλους τους σκιώδεις συζητητές και νομίζω θα λειτουργήσει καλά η συνεργασία. Αυτά για τη γενική διαδικασία. Μετά λέχθηκε ότι υπάρχουν δύο διαφορετικοί στόχοι που επιδιώκονται με την παρούσα ε, πρόταση. Αφενός καθαρότερες θάλασσες, αφετέρου αποδοτικότερες, αποτελεσματικότερες διαδικασίες στα λιμάνια. Για τις αποτελεσματικότερες διαδικασίες νομίζω ότι πιο γρήγορα το πετύχουμε αυτό παρά να καθαρίσουμε εντελώς τις θάλασσες. Αλλά αποδοτικές διαδικασίες μπορεί να εξετάσει κανείς και τι άλλες πολιτικές υπάρχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Αφενός η ενιαία θηρίδα, single window, που θα συζητηθεί σύντομα. Η ενιαία θηρίδα υπάρχει ήδη θεωρητικά όμως δεν υπάρχει ακόμα στην πράξη. Αυτό σημαίνει ότι οι διαδικασίε θα πρέπει να γίνονται ηλεκτρονικά στα λιμάνια, δηλαδή, δηλαδή ηλεκτρονικά ε, να δηλώνει το καράβι τι, όχι μόνο τι φορτίο έχει, αλλά και τι απόβλητα έχει για να παραδώσει. Αυτά να μπορούν λοιπόν να μπουν στην ενιαία θηρίδα. Για να μπορέσει να λειτουργήσει η ενιαία θηρίδα, αν μπορέσει να λειτουργήσει η ενιαία θηρίδα, θα επιταχύνει πολύ τι διαδικασίε στα λιμάνια. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αυτό αποτελεί και προπόθεση για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας. Πρέπει όμως πρωτίστως να υπάρχουν ιστοσές εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό πρέπει να διασφαλιστεί γιατί δεν υπάρχουν παντού σε όλα τα λιμάνια. Γνωρίζω ότι και πολλοί πλειοκτήτες παραπονούνται ότι ήδη στο καράβια απάνω χωρίζουν τα απόβλητα, πάνε στο λιμάνι και τα πετάνε όλα μαζί οι αρχές που τα παραλαμβάνουν. Χρειάζονται λοιπόν σωστές διαδικασίες, σωστές για την προσθέση του περιβάλλοντος να ε, ενταχθούν και στις άλλες ε, πολιτικές όπως την κυκλική οικονομία, όπως την ε, αξιοποίηση των πλαστικών απορριμμάτων και ούτω καθεξής. Έρχομαι λοιπόν τώρα στον άλλο στόχο, την καθαρότερη θάλασσα, που αποτελεί μεγίστη πρόκληση, όχι μόνο βέβαια λόγω των πλαστικών, γνωρίζουμε πρόσφατα είχαμε και την έκθεση με όλα αυτά τα πλαστικά στους ωκεανούς, όπου εγώ ήμουν πίσω από την πρόσκληση για να έλθουν να τα πούν αυτά εδώ πολλά από τα πλαστικά πέφτουν στη θάλασσα από την ξηρά, αλλά και από τα καράβια και πολύ συχνά μάλιστα και από τα αδιευτικά σκάφη. Εδώ προτάσω μία παρατήρηση. Κάτι που βρίσκω καλό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασκεί κάποια πίεση στην ΙΜΟ, στην ΑΕΜΟ, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, για να εφαρμοστεί καλύτερα και η ε, συνθήκη Μαρπόλ. Εγώ είμαι άνθρωπο ε, θετικό. Εγώ θεωρώ ότι η Μαρπόλ περιλαμβάνει πράγματα που είναι καλά για το περιβάλλον. Εάν όμω εξετάσει κανεί το παράρτημα 1 τη Μαρπόλ, βλέπει ότι επιτρέπει η Μαρπόλ να πετάγονται ορισμένα απόβλητα κατευθείαν στη θάλασσα. Αυτό δεν είναι καλό για το περιβάλλον, πρέπει να αλλάξει. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει θαύματα, ούτε και εμεί ω Ευρωβουλευτέ. Δεν μπορούμε να αναγκάσουμε όλο τον κόσμο να πάψει να κάνει τέτοια πράγματα. Αλλά μπορούμε να ασκήσουμε πίεση παίζοντα ένα ρόλο πρωτοπόρου, ώστε να αλλάξει και η Μαρπόλ. Για παράδειγμα, αδειάζουν τις δεξαμενές ε, πετρελαίου κατευθείαν στη Βόρεια Θάλασσα, αντί να περιμένουν να πάνε σε ειδικές εγκαταστάσει στο λιμάνι. Και εκεί, ε, ίσως κάπως αφελώς, πίστευα ότι το 2015 είχαμε πει μόνο 0,1% θείου στα καύσιμα τώρα έχουν πολλά καράβια συστήματα scrubber στην, στα ε, πλοία. Δεν απαγορεύεται καταρχήν να ρίξουν στη θάλασσα αυτά τα νερά τα οποία είναι μολυσμένα με θείο και με τα οποία έχουν πλύνει τις ε, έξαμενές τους. Αλλά μετά από πολλές δεκαετίες που έχει αρχίσει αυτή η, εμπορική, ε, η πρακτική, βλέπει κανείς τώρα ότι υπάρχουν μεγάλες συγκεντρώσεις θείου που δεν έχουν καμία απολύτως άλλη δικαιολογία, εκεί δηλαδή που πλησιάζουν τα καράβια στα λιμάνια, παρά μόνο αυτή, αυτόν τον καθαρισμό. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα που να λειτουργεί για την απόθεση και παραλαβή των αποβλήτων που είναι όμως, αναφέρεται για την ώρα η νομοθεσία αυτή μοναχά στα στέρεα απορρίμματα, στέρεα απόβλητα, όχι στα υγρά. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη ωστόσο στη νέα νομοθεσία. Έχω και ορισμένα άλλα ε, ζητήματα, βέβαια δεν θέλω να μονοπολίσω το μικρόφωνο, να μιλήσουν και οι άλλοι σκιώδεις εισηγητές, και άλλοι σκιώδεις εισηγητές. Ορισμένα πράγματα ήδη έχουν συζητηθεί και οι σκιώδεις εισηγητές έχουν δεχθεί επισκέψεις ε, εκπροσώπων λόμπι τα λιμάνια λένε ότι το ζήτημα είναι αν είναι σωστό να πληρώνουν εφάπαξ τα καράβια το 100% για τα απορρίμματα. Τι γίνεται όμως αν είναι hazardous waste, αν είναι δηλαδή επικίνδυνα απόβλητα, θα πρέπει να υπάρξει κάποια σταδιακή αύξηση των τελών. Θα πρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει να ληφθεί πρόνοια ώστε να μην υπάρξει κίνητρο κανένας να πετάει πλέον τα απόβλητα αυτά στη θάλασσα. Κατανοώ ότι λένε 100% καλύπτεται, επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να πετάξει κανένας πια από το καράβι τα απόβλητα στη θάλασσα, αλλά νομίζω ότι το ζήτημα αυτό πρέπει να ενταχθεί και στην κυκλική οικονομία και έχουμε στην πρόταση, στην νομοθετική πρόταση και μια πρόταση που λέει ότι εφόσον δείξει Κάποιο πολύ φιλική συμπεριφορά προς το περιβάλλον, τότε ανταμείβεται, δηλαδή πληρώνει λιγότερα εν τέλει για την ε, απόθεση των απορριμμάτων. Αν όμως γνωρίζω ότι με το τέλος που έχω καταβάλει μπορώ να αποδώσω στην ε, κατάσταση παραλαβής ο 100% των αποβλήτων δεν έχω κανένα λόγο να τα πετάξω στη θάλασσα. Επίσης, θα πρέπει να τα έχουν παραδώσει όλα τα απόβλητα πριν εγκαταλείψουν τα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολλά λιμάνια όμως σε τρίτες χώρες δεν έχουν τις εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων. Μπορεί όμως να υπάρχει και ένα πολύ σύγχρονο λιμάνι σε κάποια τρίτη χώρα, ανεξαρτήτως Brexit τώρα, το οποίο μνημονεύεται κάπου κάπου, κάπου, κάπου. Ενώ μπορεί το τελευταίο λιμάνι που ε, επισκέπτεται το καράβι στην Ευρώπη, να είναι ένα μικρό λιμάνι το οποίο δεν έχει τη σχετική κατάσταση, θα πρέπει τότε να μπορεί να, παραδώσει τα απορρίμματα στην πρώτη ε, κατάσταση που θα βρει εκτό Ευρώπη. Και τέλο, κάτι που λέχθηκε ήδη και γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το έχει πει ήδη, γιατί στι χώρε μέλη έχουν πει και το ίδιο θα έλεγα και εγώ. Υπάρχουν ήδη αλλιευτικά σκάφη τα οποία συλλέγουν απορρίμματα θα έπρεπε οι άνθρωποι και τα φέρνουν μετά στη στεριά. Δεν θα πρέπει μετά να αναγκάζονται να πληρώνουν από πάνω για να τα διαθέσουν στι εγκαταστάσει παραλαβή. Θα πρέπει αντίθετα να ανταμείβονται. Αυτά λοιπόν για την ώρα. Αναμένω με ενδιαφέρον τι προτάσει των Shadows και την περαιτέρω πορεία τη νομοθετική διαδικασία. Ευχαριστούμε. Οι εισηγητές τώρα. Η κυρία Κλούν πρώτα. Ελκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σημερινή της παρουσίαση και την εισηγήτρια βέβαια. Θέλω και εγώ να υπογραμμίσω αυτά που είπε στην αρχή, ότι ναι, θα συνεργαστούμε καλά μεταξύ μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα συμπληρωθεί ο φάκελος αυτός. Είναι μια σαφής πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ίσως να υπάρχουν κάποια στοιχεία που θα έπρεπε να συζητηθούν παρετέρω, να ζητήσουμε κάποιες αλλαγές. Συνολικά όμως το πνεύμα, η προσέγγιση της πρότασης αυτής είναι κάτι σωστό. Που λέω ότι πρέπει να μειωθούν τα απόβλητα στους ωκεανούς μας, στις θάλασσές μας. Και για να το κάνουμε αυτό πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό πρέπει να τονιστεί, να υπογραμμιστεί. Είναι καλή και συνολική αυτή η προσέγγιση. Συνεπώς, η οδηγία του 2000 σίγουρα πρέπει να ενημερωθεί και να ευθυγραμμιστεί και με την Μάρπολ, προκειμένου να μειωθεί το διοικητικό άκθος. Είμαστε υπέρ αυτού. Τώρα ασχολούμαστε πολύ με τη μείωση των πλαστικών στις θάλασσες και γενικότερα με τα πόβλητα, αλλά κυρίως με τα πλαστικά, οπότε σίγουρα θα συζητηθούν τέτοιες διατάξεις. Θέλουμε λοιπόν προστασία του θαλάσσιου χώρου και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων στους λιμένες. Αυτή είναι η στόχη και αναγνωρίζω αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν είναι όλες οι θάλασσες ίδιες, δεν είναι η ίδια αντιμετώπιση που ταιριάζει σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλα τα λιμάνια, αλλά πάντως πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα κίνητρα για να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Και να υπάρχει και ισορροπία βέβαια στις προτάσεις μας. Και να σεβόμαστε όλους τους ενδιαφερόμενους και όλους τους κλάδους. Το γεγονός ότι αυτή η απέτηση παραλαβής δεν ισχύει στα μικρά απομακρυσμένα λιμάνια είναι κάτι θετικό. Δεν έχουν και αρκετό προσωπικό για να τα ανταπεξέλθουν. Επίσης, γι' αυτό που είπε η συγκήτρια για τον προορισμό ε, σκαφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι μπορεί εκεί να πρέπει να γίνει η παράδοση, γιατί μπορεί να έχουν καλύτερες εγκαταστάσεις από ότι το τελευταίο ευρωπαϊκό λιμάνι στάσεις, όπως είπε και η συγκήτρια. Και δεδομένου του Brexit αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Έχουν πολλά και αποτελεσματικά λιμάνια που θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτήν την ε, διαδικασία. Τώρα, ότι θα πρέπει να γίνεται παράδοση σε κάθε λιμάνι Δεν νομίζω ότι πρέπει να ταλαιπωρηθούμε περισσότερο. Πρέπει να ρωτήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σε θέση όλα τα λιμάνια να ανταπεξέλθουν. Και για τη διαφοροποίηση των τελών ανάλογα με το είδος των αποβλήτων, απορριμμάτων και τα λοιπά που παραδίδονται. Όπως είπε και η συγκήτρια, μιλήσαμε με διάφορους λόμπιστς ενδιαφερόμενους και το θέμα των μικρών σκαφών κάτω από κάποιο μήκος δεν πληρώνουν αυτά τα τέλη. Θα μειωθεί το τέλος για τα μικρά αυτά σκάφη δεδομένων των δραστηριοτήτων τους και επίσης για τις εξαιρέσεις μερικές φορές τα σκάφη αναψυχής ή πολύ μικρά σκάφη θα έπρεπε να ξερούνται. Πρέπει να το δούμε και αυτό στις συζητήσεις μας. Πάντως, συνολικά, ε, όλοι αναγνωρίζουμε ότι πρέπει να πετύχουμε τους στόχους που αναφέρονται σε αυτήν την ε, πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε καρποφόρες συζητήσεις και θα συνεχίσουμε με την εισηγήτρια και τους υπόλοιπους όδες εισηγητές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Γκραπίνη, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας πω ότι με ικανοποίησαν αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και όπως και οι συνάδελφοι, έτσι και εγώ χαίρομαι. Με αυτά που είπε και η Γκεζίνε επίσης και η συνάδελφος από το ΕΛΚ. Πιστεύω ότι είμαστε στην ίδια γραμμή όλοι. Δηλαδή ξεκινάμε από τέτοιο σημείο κίνηση. Συμφωνούμε όλοι ότι μετά από 17 χρόνια η οδηγία αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί και πρέπει πολλά πράγματα να αποσαφινιστούν. Θα υπάρξουν βέβαια τροπολογίες και θα περάσουμε αρκετό χρόνο συζητώντας για το σύστημα τελών, όπως έλεγε και η Γκεζίνε. Όσον αφορά εμένα πάντως την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δεν βλέπω κίνητρα και δεν βλέπω η αρχή ορυπαίνων πληρώνει είναι εφαρμόστε. Αν όλοι πληρώνουν τα ίδια, ανεξάρτητα από τον όγκο των αποβλήτων, ε, δεν θα τηρηθεί αυτή η αρχή που λέει ορυπαίνων πληρώνει. Άρα λοιπόν πρέπει να υπάρχει μια διαφοροποίηση ανάλογα με τον όγκο των αποβλήτων. Και αυτό το τέλος, ίδιο για όλους, θα πλήξει τα μικρά σκάφη και τους μικρούς λιμένες περισσότερο. Εδώ χρειάζεται και λίγο ηθική αντιμετώπιση, δηλαδή να υπάρχει μια ηθική φορολόγηση και να υπάρχει κίνητρο ώστε να μην γίνεται η απόρριψη των αποβλήτων στη θάλασσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ίσως θα μπορούσε να μας ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα που για μένα δεν είναι σαφή. Για παράδειγμα, πώς καταλήγεται στην ιδέα του ελέγχου με το 20% γιατί όχι 30% γιατί όχι κάτι άλλο γιατί προτείνεται το 20% έπειτα ε, στα στοιχεία που συμπληρώνονται για το είδος των αποβλήτων βάσει της Μάρπολ χρειαζόμαστε και κάτι άλλο, μια ευρωπαϊκή ταξινόμηση σύμφωνα με τους δικούς μας κανόνες. Χρειάζεται ε, μια ευρωπαϊκή ταξινόμηση και αυτή να λαμβάνεται υπόψη. Τώρα γιατί η δικιά σας πρόταση δεν προτείνει τίποτα για τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα μηχανήματα λίευσης. Μα πρέπει να πάρουμε κάποια μέτρα όταν χάνεται εξοπλισμός ε, στη θάλασσα. που δεν, εξοπλισμό που δεν χρησιμοποιείται πια. Είναι σημαντικό να προχωρήσουμε σε μια οικονομία που δεν ρηπαίνει, αλλά πρέπει να συμπεριλάβουμε και τον εξοπλισμό, πιστεύω, τον αληφτικό εξοπλισμό. Ανεφερθήκατε στα πράσινα σκάφη και ελπίζω και εγώ η ομάδα μου να συμφωνήσει. Δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα, οπότε δεν ξέρω. Πάντως αυτή η αρχή ε, των πράσινων σκαφών ενθαρρύνει την ταξινόμηση των αποβλήτων πάνω στο σκάφος και μετά έτσι να παραδίδονται χωρισμένα τα απόβλητα, όπως γίνεται στις πόλεις. Και όσον αφορά το πεδίο εφαρμογή, αυτό νομίζω ότι πρέπει να επεκταθεί περισσότερο για να συμπεριλάβει και τα εσωτερικά ύδατα. Γιατί έχουμε τη θάλασσα, αλλά έχουμε και απόβλητα και στα εσωτερικά μας ύδατα. Και έχουμε πρόβλημα στον Δούναβη, για παράδειγμα, που γίνονται μεγάλες απορρίψεις και στην Μαύρη Θάλασσα και αλλού. Κάτι το οποίο φυσικά και έχει επιπτώσει... στο περιβάλλον και στα υπόγεια ύδατα. Έχοντας μιλήσει με την ομάδα μου, αφού έχω μιλήσει με την ομάδα μου, θα κάνω προτάσεις και εγώ στην εισηγήτρια και στους κοιόδης εισηγήτες. Πιστεύω ότι μπορεί να βελτιωθεί περισσότερο ακόμα αυτή η πρόταση, αλλά σίγουρα ξεκινάει από ένα πολύ καλό σημείο εκκίνησης. Και ελπίζω ότι όντως θα ολοκληρωθεί η πρόταση αυτή και θα αποφασιστεί ε, κατά τη διάρκεια της Αυστριακής Προεδρίας. Ωραία. Ο κύριος Βαντάλεν. Πέτερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ την εισηγήτρια και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Ε, στηρίζω και εγώ τους στόχους της νέας αυτής πρότασης για την μείωση των αποβλήτων ε, στη θάλασσα και να επικεντρωθούμε και στα πλαστικά. Συμφωνώ με όλα αυτά. Κανένα πρόβλημα με την προσέγγιση αυτή ως σημεία κίνηση. Όμως έχω κάποιες ερωτήσεις και ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορέσει να βοηθήσει. Πρώτα απ' όλα το θέμα της αρχής. Δηλαδή, τι χρειαζόμαστε αυτή τη νέα πρόταση. Αυτό φαίνεται λίγο τρελό, γιατί αν δούμε τι έχει γίνει στην πράξη τα τελευταία χρόνια, είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή η εφαρμογή και η διαχείριση των ε, κανόνων που ήδη έχουμε δεν είναι δυνατόν να λυθούν όλα τα προβλήματα όλε τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ακριβώ η εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την τάση πολύ γρήγορα να προτείνει νέα νομοθεσία, χωρί να έχει φροντίσει να τεθεί σε εφαρμογή ικανοποιητικά η προηγούμενη. Και με αυτό την υπερβολική νομοθετική ρύθμιση γίνεται ακόμα μεγαλύτερο μπέρδεμα και είναι ακόμα πιο δύσκολη διαχείριση των ε, κανόνων και εφαρμογή του. Οπότε, ρωτάω, η νομοθεσία που έχουμε στη διάθεσή μας μέχρι τώρα δεν ε, θα έφτανε αν όντω εφαρμοζόταν. Εγώ έτσι πιστεύω. Πέρα από αυτό το θέμα αρχής, έχω και κάποια πρακτικά ζητήματα. Διαβάζω λοιπόν το άρθρο 7 που μιλάει για την παράδοση στα λιμάνια και ότι κάποια λιμάνια ε, θα εξαιρούνται. Οπότε, εγώ ρωτάω, τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Και τι σημαίνει επαρκείς λιμανικές εγκαταστάσεις. Ποιος το ρίζει το ποιες είναι επαρκείς και ποιες δεν είναι. Γιατί τελικά ένα σωρό λιμάνια θα έρθουν και θα πούν ότι δεν έχουν επαρκείς, οπότε δεν χρειάζεται να τηρήσουν και αυτό αυτές τις διοικητικές Εμένα με εκπλήσει που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή τη δεν κάνει την ε, σύνδεση με αυτό το στοιχείο. Γιατί οι, τα λιμάνια τα οποία δεν έχουν αυτές τις εγκαταστάσεις όντως εξαιρούνται. Θα έπρεπε λοιπόν εγώ πιστεύω να το δούμε καλύτερα αυτό. Επίσης, Είμαι στην Επιτροπή Αλίας και κοιτάω λίγο και την ε, θέση του αλλιευτικού κλάδου. πολύ αλείς από πολλές χώρες, κυρίως στη Βόρεια Θάλασσα, δραστηριοποιούνται σε θελοντική ε, βάση με το πρόγραμμα Fishing for Litter, δηλαδή να μαζεύουν τα σκουπίδια στη θάλασσα. Ε, κατεστραμμένο εξοπλισμό, δίχτυα τα οποία έχουν σκιστεί και έχουν μείνει στη θάλασσα. Τα μαζεύουν λοιπόν όλα αυτά. Οπότε ρωτάω, αυτή η πρόταση δεν θα λάβει υπόψη της αυτή την ωραία πρωτοβουλία που έχουν αναλάβει πολλοί αλληλείς από πολλές χώρες μέλη. Γιατί πιστεύω ότι αυτό θα αποτελούσε ένα κίνητρο για να συμμετάσχουν ακόμα περισσότεροι σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Θα μπορούσαν δηλαδή αυτά τα απόβλητα να τα πηγαίνουν στα λιμάνια. Λοιπόν, θα ήθελα κάποια απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί ωραία είναι αυτή η πρωτοβουλία, αλλά μην ε, καταστρέψουμε υπερβάλλοντας. Πρέπει να δούμε επίσης και του ίσους όρους με τους οποίους πρέπει να εφαρμοστεί αυτή η οδηγία. Μιλήσαμε για το 100% και νομίζω ότι το ξέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τα διαφορετικά λιμάνια που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει το άρθρο 8, το οποίο λέει ότι υποχρεωτικά σε κάποιες ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να παραδίδονται τα απόβλητα. Πώς όμως θα κρυθεί αυτό. Δεν μπορούν όλα τα λιμάνια να το κάνουν αυτό. Δεν μπορούν να τα παραλάβουν και κυρίως δεν μπορούν να τα επεξεργαστούν. Ιδίως τα λιμάνια όπου έρχονται κρουαζιερόπλια. Οπότε η ερώτησή μου είναι γιατί δεν προβλέπετε λιμάνια τα οποία πρέπει να καλύψουν αυτό το κόστος να έχουν την δυνατότητα να έχουν κάποια επιδότηση, κάποια βοήθεια. Όταν ένα σκάφος φέρνει περισσότερα από ένα μέσο όρο τον οποίο θα αποφασίσουμε, τότε θα θεωρήσουμε ότι αυτό το λιμάνι δικαιούται όντως κάποια ενίσχυση. Νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό και θα ήθελα την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από αυτού. Εγώ φυσικά θα υποβάλω τροπολογία προς αυτήν την κατεύθυνση. Συνεπώς, ναι, μεν στηρίζω την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την μείωση των αποβλήτων στη θάλασσα, εννοείται. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήμουνα σε ένα παντοπολείο και όλα τα γκουράκια ήταν εκεί τυλιγμένα με πλαστικό. Πώς θα μειωθούν τα πλαστικά έτσι. Λοιπόν, πρέπει να συζητήσουμε και τέλος θέλω να ρωτήσω και την εισηγήτρια κάτι. Αν έχω διαβάσει καλά, πρέπει μέσα σε 6 εβδομάδες μέχρι τις 18 Ιουλίου, παρόλο που δεν έχουμε κείμενο, να υποβάλουμε τροπολογίες. Πώς θα γίνει αυτό. 18 Ιουλίου, μα τότε αρχίζουν οι καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε ρωτάω, μπορούμε να το λάβουμε όψη μας αυτό. ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Βαντάλε. Για τους πράσινους, Τέιλορ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την Επιτροπή και την εισηγήτρια. Εμείς ε, συμφωνούμε με την πρόταση ότι πρέπει να αντικατασταθεί η παλιά οδηγία και να ξεκινήσουμε από την αρχή. Και διαπιστώνω πως υπάρχει μια ευρύτερη κοινή βούληση για βελτιώσεις στις ε, λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής, αλλά και υπέρ των πρωτοβουλειών μείωσης των αποβλήτων. Μια εβδομάδα όπου είδαμε στην Ταϊλάνδη το θάνατο μιας ε, φάλαινας που είχε καταπιεί ε, από ό,τι φαίνεται 80 πλαστικές σακούλες. Ε, αυτές ήταν στο, στο μάχη της και τη, δεν την άφηναν πια να τραφεί. Αυτό καταδεικνύει πού βρισκόμαστε. Κατά τη γνώμη μου, λοιπόν, όποιος κανονισμός υπάρχει αυτή τη στιγμή, σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί. να μην επιτρέπεται να συνεχίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Πολύ θα ήθελα λοιπόν να τα κίνητρα που περιγράφηκαν για την ε, αύξηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων στα λιμάνια να συνοδεύονται ίσως και από βελτιωμένη επιβολή. Δεν έχω ιδέα πώς θα γίνει αυτό, ποιες είναι οι τεχνικές δυνατότητες, αλλά μπορούμε ίσως να παρακολουθούμε τι γίνεται με το σύστημα το δορυφορικό για την ασφαλή θάλασσα. Υπάρχει ένα τέτοιο δίκτυο και να εντοπίζουμε αν γίνονται και αν υπάρχουν εκπομπές, ε, μάλλον ρήψεις στη θάλασσα και ίσως και να, έτσι να προβούμε σε δράσεις κατά των ιδιοκτητών των σκαφών ή του καπετάνιου, του πλοίαρχου. Το καλύτερο είναι να υπάρχει αυτός ο κατάσκοπος στο εξ ουρανού, ε, που θα είναι πάντα στο μυαλό των αρμόδιων ώστε να μην ρίχνουν τα θάλασσα. Η, η θάλασσά μας καλύπτει το 70% του πλανήτη. Πρέπει λοιπόν να την προσέχουμε και όχι να συνεχίζουμε να τη ρηπαίνουμε με θείο, ε, απόβλητα, πλαστικά, αλλά να κάνουμε πραγματικά το μέσα στον χειρισμό του προβλήματος. Σίγουρα εμείς οι πράσινοι θέλουμε να συνεργαστούμε με τους υπόλοιπους σκιώδεις για να αναπτύξουμε κάτι που θα μας κάνει περήφανος και θα σημάνει τη διαφορά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Τέιλορ Η κυρία Γκοζάλες Πένιας. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την Επιτροπή το γεγονός ότι ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία που είναι τόσο σημαντική σε μια φάση όπου μπορούμε να μιλήσουμε σχεδόν για το boom των θαλάσσιων μεταφορών, όχι μόνο για τον τουρισμό αλλά και για τη μεταφορά εμπορευμάτων ε, σε διεθνές επίπεδο είναι πολύ σημαντικό και ευχαριστώ και την εισηγήτρια με την ευκαιρία και για την προσπάθεια της ε, στην Ήπειρό στην Ευρωπαϊκή που είναι στην ουσία σαν μια τεράστια χερσόνησος και έχει τεράστια ιστορία στη θάλασσα ε, θα πρέπει να αναλάβουμε την ευθύνη της αποσταθεροποίησης και της βλάβης στον πλανήτη με αυτήν μας την θαλάσσια δραστηριότητα. Είναι ένα καθήκον, μια υποχρέωσή μας, ε, θα έλεγα ακόμα και ηθική ε, και αυτό ήδη γίνεται με την Μαρπόλ και θέλω να πω και για τη χώρα μου που πάλι είναι ακόμα ένα ε, κομμάτι, μια χερσόνησος της Επίρου ε, ε, θέλουμε να διατηρήσουμε τις ακτές και τις παραλίες μας, ε, τη θάλασσά μας και να προστατεύσουμε και το μέλλον της τουριστικής δραστηριότητας. Μπορεί να μιλήσει κανείς για την Ισπανία, για την Ιταλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία, την ε, Γαλλία, την, την Φιλανδία, τη Σουηδία κτλ. Χώρες ε, όπου τα νερά τους δεν αξίζουν τόσα σκουπίδια τα οποία αφήνουμε πίσω μας επειδή δεν είμαστε αρκετά διορατική. Ε, συμφωνούμε λοιπόν με αυτή την οδηγία. Υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία όπως ας πούμε η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής ή ότι τα τέλη εξαρτώνται από τον όγκο των ε, ρήπων που παραδίδονται, ε, που ξεφορτώνονται στα λιμάνια, δηλαδή ένα σημαντικό κίνητρο για να πετιούνται τα σκουπίδια στα λιμάνια και όχι ε, στην ανοιχτή θάλασσα. Υπάρχουν όμως και σημεία που πρέπει να δουλευτούν περισσότερο. Καταρχάς να την υποχρέωση και τους στόχους κατάρτισης για το ναυτικό προσωπικό, όχι μόνο αυτούς που χειρίζονται τα απόβλητα, αλλά και όλους εκείνους τους λιμενικούς εργαζόμενους ε, που μπορεί να εργάζονται στις εγκαταστάσεις και χειρίζονται τους όγκους αποβλήτων που ε, ξεφορτώνονται εκεί. Έπειτα, κύκλος επιθεωρήσεων. Θα πρέπει εκεί να περιλαμβάνονται και τυχαίοι έλεγχοι και τυχαίες επιθεωρήσεις, ε, απροειδοποίητες δηλαδή. Επίσης, ε, να περιλαμβάνουμε ε, μάλλον να καταγράφουμε και τις κυρώσεις που επιβάλλουν τα κάτι μελη για τα αδικήματα κατά της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος. Αυτά ε, γενικά φυσικά και είμαστε έτοιμοι να ε, συνεργαστούμε για την εμβάθυνση σε αυτή την πρόταση. Ευχαριστώ. Σκιώδης ε, ολοκλήρωσαν οι δύο με τρία λεπτά υπόλοιποι συνάδελφοι. Κυρία Φώστερ πρώτα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εσάς και Ζήνε δεν είμαι εκ των σχεδόν εισηγητών, αλλά έχω λίγα σύντομα σχόλια. Ανησυχούμε πολύ για την ε, διάθεση των αποβλήτων. Από τότε που ταξιδεύω έχω δει άπειρα απόβλητα στις θάλασσες και όχι καράβια μόνο. Και ο Πίτερ Βαντάλεν έθεσε το θέμα της επιβολής της νομοθεσίας Τη υφιστάμενη Νομοθεσία, είτε εθνικής είτε ευρωπαϊκής για θέματα περιβάλλοντος. Τώρα για το, για το σύστημα των τελών. Πρέπει να συνδεθεί με τους επιδιωκόμενους στόχους. Ορισμένα σκάφη δεν έχουν επικίνδυνα απόβλητα. Αυτό που μπορεί να συμβεί δηλαδή τελικά είναι ότι ορισμένα πλοία που ε, δεν διαθέτουν τέτοιου είδου απόβλητα μπορεί τελικώ ή έχουν πολύ μικρότερο ποσοστό να πληρώνουν δυσανάλογα υψηλά τέλη. Και τότε μπαίνουμε στο θέμα του ο ρηπαίνων πληρώνει. Τώρα, για την διάθεση των αποβλήτων, εάν βέβαια αυτά είναι υγρά απόβλητα, αυτά μετρώνται όπως μετρώνται τα απόβλητα. Αλλά για στερεά απόβλητα αυτό γίνεται με κυβικά μέτρα. Και αυτό γίνεται με, με, με το μάτι περίπου, δηλαδή, ε, αλλά δεν είναι ακριβής. Πώς θα αποδώσουν τα συστήματα αυτά. Το άλλο είναι το πού διατίθενται τα απόβλητα ή απορρίμματα. Όταν τώρα κάποια δεξαμενή ή κάτι άλλο έχει γεμίσει, το αφαιρούν από το σκάφος. Αλλά πρέπει όμως να υπάρχουν απαιτήσει και για τον εργολήπτη που θα κάνει την παραλαβή. Θα πρέπει να είναι υπόλογος και για το τελευταίο απόβλητο. Αυτό όμως σημαίνει τεράστια γραφειοκρατία και κόστος και δεν μας εξυπηρετεί οι ε, χώρες μέλη, τα λιμάνια, θα πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν να παραλάβουν τα απόβλητα και να τα διαθέσουν όπως πρέπει κλπ. έχουν άδεια λειτουργία όπως προβλέπεται από τον νόμο και να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Και αυτό που είπε ο Keith Taylor είναι σημαντικό. Παρακολούθηση από δορυφόρους και η χνηλασιμότητα. Να δούμε δηλαδή ποιος είναι ο υπεύθυνο για την απόρριψη των αποβλήτων στη θάλασσα. Κατά τα λοιπά νομίζω ότι τα έχουν πει όλες οι συναδελφοί μου, αλλά πρέπει να προσέξουμε πολύ τις προτάσεις που κάνει η Κομισιόν. Ευχαριστώ κύριε Φώστερο, κύριος Κράμερ. Ευχαριστώ πολύ και την Κομισιόν και την εισηγήτρια και τους υπολείπους για τις παρεμβάσεις. Έρχομαι σε κάτι που είπε ο Πέτερ Βαντάλεν. Εάν δεν ελέγχεται η εφαρμογή ενός νόμου, τότε είναι περιττός ο νόμος. Περί αυτού πρόκειται. Βεβαίω αντιλαμβάνομαι ότι έχει τι για την εφαρμογή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τι κάνουν οι χώρε μέλη. Θα ήθελα να μάθω από την Επιτροπή αν έχει μιλήσει με τις χώρε μέλη, πώ αντέδρασαν οι χώρε μέλη, ιδίω πώς αντιδρούν στο ερώτημα του ελέγχου. Μιλήσαμε για το θείο στο αργό πετρέλαιο. Είπαμε ότι πρέπει να μειωθεί στο 1%. Γίνεται έλεγχος. Πώς γίνεται ο έλεγχος. Είχαμε πει από την αρχή καλύτερα θα ήταν Είχαμε πει από την αρχή να μην υπάρχει καν να χρησιμοποιείται δίζελ. Όμως το αργό πετρέλαιο είναι πολύ φθηνότερο από το δίζελ και τελικώ χρησιμοποιείται. Η ερώτησή μου είναι πώ γίνεται ο έλεγχο Και Ζήνε γνωρίζει, το έχουμε συζητήσει το ζήτημα αυτό, μέσα στα απόβλητα, τα απόβλητα μάλλον, τα πετάνε στη θάλασσα τα καράβια και 5 και 10 και 20 χιλιόμετρα πριν από το λιμάνι. Και δεν χρειάζεται να πληρώσουν τέλη όταν φτάνουν στο λιμάνι. Αν αυτά τα πράγματα δεν ελεγχθούν αυστηρότατα και να τιμωρηθούν αυστηρότατα, δηλαδή ο κίνδυνος του προστίμου να είναι τόσο υψηλός που να τους αποθαρρύνει. Απολύτως. Αυτά. Και θα ήθελα να μάθω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι εμπειρίες έχει από τη συζητήση με τις χώρες μέλη. Σας ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω την εκπρόσωπο της Επιτροπής να απαντήσει σε λίγα λεπτά στις ερωτήσεις της ε, εισηγήτριας καθώς και των υπολείπων ευρωβουλευτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια και τα άλλα μέλη της Επιτροπής σας που έλαβαν το λόγο και συζήτησαν το θέμα. Να αρχίσω με ένα κάπως ασυνήθιστο τρόπο. Πολλοί από εσά επενέσατε την πρόταση, ότι είπατε ότι είναι σαφής και λεπτομερής. Οι έπαινοι αξίζουν στην κοπέλα που κάθεται αριστερά μου, που έκανε όλη τη δουλειά, την Άννα Μπορένκο. Οποιαδήποτε λεπτομέρεια τη γνωρίζει απ' έξω. Δεν θα μπορέσω όμως να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας λόγω χρόνου. Αλλά είμαι ανα πάσα στιγμή στη διάθεσή σας για να απαντήσουμε και σε άλλα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, για λίγα λεπτά επιτρέψτε μου, διότι όλες οι ερωτήσεις σα βελτιώνουν τη συζήτηση και αυτή που θα γίνει στις επόμενες συνεδριάσεις. Θα, τα πω λίγο, θα απαντήσω λίγο ανακατεμένα. Πάντω μια ερώτηση που έγινε από τον κύριο Βαντάλεν, αν δεν αρκεί να εφαρμόσουμε τι υφιστάμενε νομοθετικέ διατάξει. Ένα από του λόγου που θεωρήσαμε ότι πρέπει να αναθεωρηθεί είναι διότι έχει αλλάξει η παγκόσμια τάξη. Η Μαρπόλ αναβαθμίστηκε, η σύμβαση Μαρπόλ. Είναι πιο προωθημένη από αυτήν που είχαμε πριν. Αντιμετωπίζαμε λοιπόν μια κατάσταση όπου αφενό τα σκάφη δεν επιτρέπεται να πετούν στη θάλασσα κάποια είδη απορριμμάτων, δεν έχουμε όμω αρμόζουσε λύσει που να επιτρέπουν να διατεθούν τα απορρίμματα αυτά κάπου. Άρα τελικά σιωπηρό θα αποδεχόμασταν ότι θα πέταγαν τελικώ τα απορρίμματα στη θάλασσα κοντά στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έρχομαι σε ένα άλλο ερώτημα που θέσατε ορισμένοι εξημών. Εάν δηλαδή τα απορρίμματα πρέπει να διατίθενται σε κάθε λιμάνι, εάν τα λιμάνια έχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις παραλαβής. Αυτό είναι το βασικό σημείο της οδηγίας. Δεν χρειάζεται να είναι σε κάθε λιμάνι. Προβλέπονται λύσεις στην οδηγία που επιτρέπουν εξαιρέσει από την παράδοση σε κάθε λιμάνι. Όμως, έχει και ένα καθαρό μήνυμα η οδηγία. Τα λιμάνια θα πρέπει να είναι έτοιμα να παραλάβουν τα απορρίμματα στην βάση του συνήθους φόρτου εργασία, του, δηλαδή του συνήθους αριθμού πλοίων που υποδέχονται. Είναι κάτι που δεν μπορεί να σχεδιαστεί, δεν μπορεί να προγραμματιστεί εκ των προτέρων. Και γι' αυτό πρέπει να προγραμματίσουν τα λιμάνια από πριν πώς θα διαχειριστούν τα παραδιδόμενα απορρίμματα, απόβλητα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι σημαντικό για την ορθή εφαρμογή και λειτουργία τη οδηγία. Και γνωρίζω ότι πολλά λιμάνια, βεβαίω έχουμε συζητήσει μαζί τους, και στην δημόσια διαβούλευση, αλλά και αυτή τη στιγμή προωθήθηκε η οδηγία. Αλλά νομίζω ότι εδώ κρύβεται κάποια παρανόηση. Δεν θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι τα λιμάνια θα μπορούν να πούν γνωρίζοντας ποια καράβια θα έρθουν. Δεν είμαστε έτοιμα να υποδεχθούμε, διότι τότε είναι μια ευθεία πρόσκληση προς τους ε, εφοπλιστές, πλειοκτήτες και λοιπούς να τα πετάξουν στη θάλασσα. Στο ίδιο πλαίσιο, η ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών θα βοηθήσει πάρα πολύ. Έγινε και μια ερώτηση σχετικά με την υποχρέωση κοινοποίηση, reporting obligation. Και είπε η κυρία Φώστερ ότι είναι κάπως ε, δυσκίνητη. Έχουμε όμως ήδη ηλεκτρονικό τρόπο advanced waste notification, κοινοποίησης δηλαδή εκ των προτέρων που κινείται ηλεκτρονικά και στην παρούσα πρόταση αναθεώρησης για την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας δηλαδή, αυτό θα προχωρήσει, θα εναρμονιστεί δηλαδή η κοινοποίηση αυτή, θα διευκολυνθεί και άλλο η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ διαφόρων λιμανιών, ώστε να εξασφαλιστεί ότι το σκάφο που έχει εγκαταλείψει ένα ευρωπαϊκό λιμάνι, τι ακριβώ έχει κάνει και ποια είναι η υποχρέωσή του απέναντι στο επόμενο λιμάνι που θα πιάσει. Πολλοί από εσά άλλωστε είπατε σχετικά με τα τέλη και ιδίως αν είναι δίκαιο να εφαρμοστεί αυτό το σύστημα έμεσων τελών. Εμείς εξετάσαμε προσεκτικά το σύστημα. Στη βάση του, εάν επιλέξουμε την προσέγγιση του άμεσου τέλους, δηλαδή πληρώνει το καράβι ακριβώς αυτά που, για αυτά που παραδίδει. Δυστυχώς, ε, έτσι όπως λειτουργεί ο κόσμος, είναι ενθάρρυνση για ορισμένους είτε να μην παραδώσουν καθόλου απορρίμματα και απόβλητα, είτε να μην είναι πάντοτε ειλικρινείς στην ανακοίνωση του τι παραδίδουν. Από την άλλη μεριά, απλή δήλωση ότι πληρώνει ούτως ή άλλως, είτε παραδώσεις απορρίμματα ή όχι, είναι ένα καθαρό κίνητρο για να παραδίδουν τα απορρίμματα όταν φτάνουν στα λιμάνια δεν θα είναι το ίδιο τέλο λόγω του μεγέθου. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι τα μικρά σκάφη θα πληρώνουν περισσότερο μόνο επειδή είναι μικρότερα. Όμως το σύστημα των έμεσων τελών είναι αποτελεσματικό και έχουμε προβλέψει και την εξαίρεση με το 100% τέλους για απορρίμματα, για σκουπίδια εν προκειμένου δηλαδή. Η οδηγία προβλέπει και το δικαίωμα παράδοσης ο Πρόεδρος. Σας παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Σας δώσαμε πολύ χρόνο πριν για να παρουσιάσετε το θέμα και σιγά σιγά αρχίζουμε να σημειώνουμε καθυστέρηση. Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας. Πρόσωπος της Κομισιόν. Λυπούμε πολύ. Ε, ανησυχούσα και εγώ λιγάκι ότι ίσως παρασυρθώ και μιλήσω παραπάνω. Αλλά είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε λεπτομερή συζήτηση με οποιοδήποτε μέλος της Επιτροπής σας. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ, διότι νομίζω ότι είπα τα περισσότερα. Ο Πρόεδρος διακόπτηκε πάλι. Ευχαριστώ. Θα μας παρουσιάσει την έκθεση στις 10 Ιουλίου η Γκεζίνε με προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 18 Ιουλίου αυτό θα επιβεβαιωθεί ακόμη. Η δε ψηφοφορία προβλέπεται στις 9 Δεκάτου, Οκτωβρίου δηλαδή. Και όπως είπε η εισηγήτρια, ελπίζουμε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την προσπάθεια σε συνεργασία με το Συμβούλιο πριν από την ολοκλήρωση της κοινοβουλευτικής θητείας. Αν έχετε κάτι να, πει ακόμα, να πείτε ακόμα, Γκεζίνε, θα είμαι συντομοτάτη, διότι ε, πράγματι έχουμε κάποια καθυστέρηση. Τα έχουμε θίξει όλα ένα μόνο για το χρονοδιάγραμμα. Διότι κάποιο είπε ότι είναι υπερβολικά φιλόδοξο. Εγώ θεωρώ ότι θα τα επιτύχουμε. Θα το πετύχουμε. Θα σα τα υποβάλω στα αγγλικά την επόμενη εβδομάδα. Δεν είναι και τόσο μεγάλο μακροσκελέ δηλαδή το νομοθέτημα. Οτιδήποτε άλλο για τι λεπτομέρειε, όλα αυτά που είπατε τα έχω σημειώσει. Και πολύ καλά τα συζητήσαμε. Ευχαριστώ. Ε, Ωραία. Ε, εντάξει, ευχαριστούμε. Και συμφωνούμε. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη θα συγκεντρώσω τα σημεία 5 και 6 μαζί, έτσι, γιατί πρόκειται για σημεία που είναι συμπληρωματικά μεταξύ τους και έχουν και τον ίδιο εισηγητή και τους ίδιους σκιώδεις εισηγητές. Οπότε θα τα εξετάσουμε από κοινού. Πρόκειται λοιπόν για την ε, Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών Ευρωπαϊκής Κοινότητας Καναδά και πρόκειται και για τη Συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της για να λεφθεί υπόψη προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ασής που είναι και η συγητής και μετά θα ακούσουμε και τους κοιόδης συγητές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Συμφωνία Αεροπορικών Μεταφορών που σήμερα συζητάμε ήδη έχει βρει συνένεση από το σώμα σε δύο συνεδριάσεις και ε, θα ισχύσει μετά από την υπογραφή του. Τώρα χρειάζεται να το συζητήσουμε εδώ γιατί χρειάζεται μετά από την απόφαση μάλλον του 10 διότι η διαδικασία που ακολουθήθηκε και δεν ήταν η σωστή σύμφωνα με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ο στόχος είναι η δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς αεροπορικών μεταφορών ανάμεσα στην Ένωση και το Καναδά όπου τα κεφάλαια θα κυκλοφορούν ελεύθερα και οι αεροπορικές εταιρείε οι ευρωπαϊκέ και οι καναδικέ θα μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίε χωρί προσκόμματα και στι εσωτερικέ αγορέ ε, των ΜΕ και των ΔΕ. Έτσι μετατρέπεται η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα παγκόσμιο φορέα ε, στη συνεργασία με τον Καναδά. Ε, πρέπει λοιπόν να ανοίξει η αγορά και αυτό θα γίνει σε τέσσερα στάδια. Το πρώτο ε, σημαίνει ε, συνεργασία και για τις ασφαλιστικές, στην ασφάλεια και για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων και για την ε, μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των αεροπορικών μεταφορών. Γι' αυτό και δεν μπορώ παρά να συστήσω την έγκριση αυτού, αυτής της συμφωνίας. Απόλυτα συνδέεται με αυτό και το δεύτερο θέμα και έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι ένα πρωτόκολλο που προβλέπει ε, να επιτρέψει στην Κροατία που έχει εισχωρήσει φυσικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει σε και εκείνη σε αυτή τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Καναδά και φυσικά σας προτείνω να το υπερψηφίσουμε. Ευχαριστούμε κύριε Ασής και τώρα το λόγο θα λάβουν οι σκιώδες εισηγητές που ασχολούνται και εκείνοι και με τα δύο θέματα ταυτόχρονα. Η κυρία Άκλουν για τους δύο σκιώθεις. Ευχαριστώ. Εκ μέρους της κυρίας Τέλη θα μιλήσω, που είναι σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ βέβαια τον εισηγητή για την παρουσίασή του, για το περί πρόκειται. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα. Συμφωνούμε απόλυτα βέβαια με την πρότασή του. Ξέρουμε ότι ο Καναδάς είναι πολύ βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτή η συμφωνία για τις αεροπορικές μεταφορές είναι πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά, το έχει συζητήσει, το ξέρετε κι εσείς και φυσικά και είμαστε υπέρ. Το ΕΛΚ λοιπόν σαφώς και είναι υπέρ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή για την πρότασή του λοιπόν και για την παρουσίαση που μας έκανε σήμερα το πρωί. Όλα αυτά εκ μέρους της κυρίας Ντέλη. Ευχαριστούμε κυρία Κλούν. Και κυρία Φώστερ. Και εγώ πολύ σύντομα ευχαριστώ πολύ τον εισηγητή, ο οποίος παρουσίασε με σαφήνεια τις δύο τεχνικές προσαρμογές. Πολύ σημαντική αυτή η τεχνική συμφωνία. Το ECR δεν έχει να προσθέσει τίποτα άλλο. Πρέπει να προχωρήσουμε. Ωραία, κύριος Ράντος. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Άλντε επίσης θα στηρίξει και τις δύο αυτές συμφωνίες. Ελπίζουμε ότι μετά από 7 χρόνια που ψηφίστηκε για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αυτό το θέμα. Το επόμενο στάδιο ελευθέρωσης των ε, συναλλαγών σε αυτό το κλάδο με τον Καναδά θα προχωρήσει και θα επιταχυνθεί μάλιστα. Αυτό είναι προς το συμφέρον των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά. Όσον αφορά το πρωτόκολλο για την προσχώρηση της Κροατίας, το πρωτόκολλο αυτό δεν αλλάζει τη βασική συμφωνία. Η Κροατία δεν είχε προηγουμένως συμφωνίες με τον Καναδά, οπότε οι φιλελεύθεροι θα στηρίξουν τη συμφωνία αυτή. Ευχαριστούμε κύριε Ράντος, ο κύριος Τέιλορ. Σύντομα και εγώ ε, ευχαριστώ. Μας ικανοποιεί και η μία και η άλλη πρόταση. Θα τη στηρίξουμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε που ήσασταν και σύντομο. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, Γκάιλ, εσείς κύριε Γκάιλ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Και εγώ θα είμαι σύντομος. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την εξαίρετη έκθεση. Όπως είπε και η κυρία Φώστερ, πρόκειται για μια τεχνική προσαρμογή των προηγούμενων προτάσεων. Και όπως είπε και ο εισηγητής, η Συμφωνία Μεταφορών Ευρωπαϊκή Ένωσης ε, Καναδά είναι μια από τις πιο σημαντικές και πιο φιλόδοξες που έχουμε υπογράψει ποτέ. Ο Καναδάς είναι μια από τις μεγαλύτερες αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με πάνω από 11 εκατομμύρια επιβάτες που πετούν από τον Καναδά στην Ευρώπη και του Μπαλιν. Είδαμε ότι η συμφωνία αυτή άρχισε να εφαρμόζεται από το 2009 που γράφηκε για πρώτη φορά. Είδαμε ότι υπάρχουν οικονομικά ωφέλη από τη συμφωνία ήδη όπως αναμενόταν και το βλέπουμε αυτό και από άλλες συμφωνίες μεταφορών. Έχουμε αύξηση 25% των επιβατών, 40% περισσότερες διαδρομές μεταξύ Καναδά και Ευρωπαϊκής Ένωσης, 18 επιπλέον πόλεις και χάρη σε αυτόν τον αυξανόμενο ανταγωνισμό διαπιστώνουμε ότι υπάρχει και μείωση κατά μέσο όρο στις τιμές των εισιτηρίων για τη διαδρομή αυτή, 220 ευρώ ανά εισιτήριο κατά μεσόρο. Κάτι το οποίο είναι σημαντικό και έχει οδηγήσει σε οικονομικά ωφέλη της τάξης των 2,5 δισεκατομμυρίων από το 2009 μέχρι τώρα. Οπότε ευχαριστώ πολύ για την σύσταση αυτή, για σύμφωνη γνώμη, προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία αυτή και να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι και η Κροατία έχει υπογράψει τη συμφωνία αυτή ε, προσχωρώντας την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο εισηγητή και πάλι για να ολοκληρώσει. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω του συναδέλφου για τα όσα είπαν και για τις παρατηρήσεις τους και να ευχαριστήσω και τον εκπρόσωπο της Επίτροπή. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σίγητα. Υπενθυμίζω ότι η προθεσμία για υποβολή τροπολογιών ή της γιατί δεν μπορούν να υπάρξουν άλλες τροπολογίες. Η μόνη τροπολογία που μπορεί να υπάρξει είναι διαγραφής άρνησης. Και για τις δύο εκθέσεις είναι μέχρι τις 13 Ιουνίου, 13 Ιουνίου στις 12 το μεσημέρι. Και περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης τώρα. Α, ήρθε πρόεδρος, οπότε εγώ απολύομαι. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο Λυρικέ. Κάτι έκτακτο μου συνέβη σήμερα το πρωί και γι' αυτό δεν μπόρεσα να έρθω έγκαιρα. Λοιπόν, συνεχίζουμε και είμαστε στο σημείο 7. Ανάπτυξη υποδομών για αναλλακτικά καύσιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ώρα για δράση. Η συγκητής μας είναι ο κύριος Ισμαήλ Ερτούκ. Καλημέρα. Ισμαήλ Ερτουκ. Σας δίνω το λόγο και μετά θα συζητήσουμε με τους Κιώδης και θα δώσω βέβαια το λόγο ξανά σε εσά, αφού προηγουμένω έχει μιλήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λοιπόν, σα ακούμε. Καλημέρα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, σύντομη παρουσία της εκθέσεως. Όλοι εδώ έχουμε πείρα και γνωρίζουμε ότι οι μεταφορές είναι ο τομέας εκείνος που έχει αυξήσει τις εκπομπές από το 1990 και μετά σαφέστατα. Και αν εξετάσουμε τα νούμερα θα δούμε ότι το 1 τρίτο ή στο 1 τέταρτο όλων των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακου προέρχονται από τις μεταφορές. Και πάλι από αυτό το ποσοστό περίπου τα 3 τέταρτα προέρχονται από τις οδικές μεταφορές. Και επειδή θα πρέπει να παίρνουμε σοβαρά τους στόχους του Παρισιού, θα πρέπει μέχρι το 2050 να αφαιρέσουμε τα καυσαέρια, δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με εκπομπή καυσαερίων του άνθρακος από τις μεταφορές. Αυτό έχει και οικονομικό χαρακτήρα. Το 94% της ενέργειας της μεταφορές προέρχεται από πετρέλαιο. Και από αυτά τα 94, τα 90% εισάγονται. Δηλαδή, κατά δισεκατομμύρια πληρώνουμε, δισεκατομμύρια ευρώ πληρώνουμε κάθε χρόνο σε χώρες οι οποίες δεν είναι απαραίτητα και σταθερές. Τι μπορεί να κάνει κανείς λοιπόν στις οδικές μεταφορές. Υπάρχουν πλήρωνες δυνατότητες. Έχω σημειώσει τις τρεις πιο σημαντικές. Αφενός χρειαζόμαστε ένα model shift, μια αλλαγή ε, προτύπου κυρίως για τις μεταφορές αγαθών, να μετακινηθούν δηλαδή στον σιδηρόδρομο και στη, στην εσωτερική ναυσιπλοεία. Δεύτερον, γενικά ισχύει πάλι και είναι σημαντικό να υπάρξει μείωση συνολικά των μεταφορών. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν επενδύσουμε περισσότερο σε τρόπους όπως ride sharing, δηλαδή μοίρασμα αυτοκινήτων κλπ. και κυρίως βέβαια να προωθήσουμε τι δημόσιες μεταφορές. Εν τέλει και περί αυτού πρόκειται ιδίω στην παρούσα έκθεση, πρέπει να φροντίσουμε ε, να δώσουμε ε, όθηση σε εναλλακτικέ μεθόδους και ιδίω για τις τελευταίε εναλλακτικέ μεθόδους. Δηλαδή εκεί έχουμε ένα σοβαρό έλλειμμα σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη υποδομή για εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια. Έχουμε και άλλο έλλειμμα σε ό,τι αφορά την εισαγωγή στην αγορά των σχετικών οχημάτων και εκεί υπάρχει μεγάλη υστέρηση που πρέπει να αντιμετωπιστεί, κάτι το οποίο θα μπορέσει να γίνει μόνο εφόσον οι κατασκευαστές αφενός προσφέρουν νέα μοντέλα, τα οποία όμως να μπορεί να τα πληρώσει κανείς, και δεύτερο, αν καταφέρουμε να προωθήσουμε περισσότερο την προώθηση ανεφοδιασμού των ηλεκτρικών οχημάτων. Το 2014, όσοι ήσασταν ήδη στο Ευρωκοινοβούλιο θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει ένα σχέδιο οδηγίας την 94 του 2014 οδηγία η οποία προέβλεπε και ποσοτικά μετρήσιμους στόχους για την ανάπτυξη της υποδομής ανεφοδιασμού. Δυστυχώς αυτή η σωστή προσέγγιση δεν κατέληξε πουθενά, διότι το τροπήλησαν οι χώρες μέλη στο Συμβούλιο Υπουργών. Με αποτέλεσμα να καταλήξουμε σε ένα αποδυναμωμένο συμβασμό που προέβλεπε εθνικά σχέδια πλαίσια, όπου τελικώς διαπιστώθηκε ότι κάποιοι οικειοθελείς εθελοντικοί στόχοι που ε, είχαν επαφεθεί στις ε, χώρες μέλη δεν εξεπληρώθησαν. Γι' αυτό, αυτό που ζητώ εγώ τώρα είναι η οδηγία αυτή, επειδή τελικώ δεν επέτυχε το στόχο της, να αναθεωρηθεί το συντομότερο δυνατό. Να καταργηθεί το σύστημα των εθελοντικών στόχων σε εθνικά πλαίσια σχέδια διότι δεν απέδωσαν τίποτα και χάσαμε και τέσσερα χρόνια. Οι χώρες μέλη βεβαίως έχουν διαφορετικά επίπεδα φιλοδοξίας για το θέμα αυτό. Είναι απαραίτητο να σημειωθεί αυτό. Πάντως έχουμε πολύ, υστερούμε πολύ απέναντι και στις χαμηλότερες προσδοκίες. Χρειάζονται λοιπόν φιλοδοξότεροι στόχοι, πρέπει να επαναφερθούν οι στόχοι αυτοί μέσω της νέας οδηγίας και θα πρέπει να διδαχθούμε και από τα όσα έγιναν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, διότι δεν αρκούν τα σχεδια τεν τεν-τι. Χρειάζεται να δημιουργηθούν κόμβοι και περιφερειακοί και διαπεριφερειακοί και όπως είπα δίκτυα υποδομών ανεφοδιασμού κλπ. Αυτά, μάλλον την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλει να την επενέσει κανείς διότι προβλέπει ήδη 800 εκατομμύρια ευρώ για τους ε, σκοπούς αυτούς. Δυστυχώς αλλά σε αυτό δεν φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το υπολογιζόμενο αναγκαίο κόστος είναι της τάξης των 22 δισεκατομμυρίων, οπότε τα 800 εκατομμύρια είναι σταγόνεν το ωκεανό. Επειδή μιλούμε εδώ ωστόσο για δημόσια δίκτυα ανεφοδιασμού, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από ένα European Clean Mobility Fund, ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Καθαρής Κινητικότητας. Αυτό το ταμείο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί κατά 90% από τους ενδιαφερομένους και αυτούς που θα το χρησιμοποιήσουν στο μέλλον, από τις βιομηχανίες, αφενός δηλαδή οι κατασκευαστές αυτοκινήτων, οι προμηθευτές και αυτοί που προμηθεύουν ενέργεια, τα τελευταία 10% θα πρέπει να τα καταβάλουμε εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Το, το πώς θα διαμορφωθεί αυτό αυτό είναι ζήτημα ιδίω τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έχει την σχετική εμπειρογνωσία. Ωστόσο, νομίζω ότι ένα πράγμα έχει αποδειχθεί τα τελευταία χρόνια, δηλαδή ότι η διαδικασία όπως τη χρησιμοποίησαμε στην ΣΕΦ, διευκόλυνση συνδέοντα στην Ευρώπη. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο ξεκινά από τα κράτη και νομίζω ότι ήταν και ευφυής η απόφαση που λήφθηκε. Δηλαδή, να πει ως άξονας, ως κόμβος, ειδικό οργανισμός ο οποίος συνδέει τις προσπάθειες των χωρών μελών. Και εδώ μπορεί να γίνει το ίδιο. Θα επιτευχθεί όμως μόνο εάν προσφέρουμε εύκολη προσέγγιση σε χρηματοδότηση Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων για τους κατασκευαστές. Θα πρέπει να εξετάσουμε και πάλι ποιε είναι οι εναλλακτικέ ε, μέθοδοι ή οι εναλλακτικέ αυτέ ενέργειε. Και εν προκειμένου, κατά τη γνώμη μου, θα είναι κρίσιμο να εξεταστεί και η διαδικασία υδρογόνου και να προωθηθεί η σχετική υποδομή. Βέβαια, πρόκειται για έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας. Άρα, η έκθεσή της είναι περιορισμένη. Γι' αυτό και περιορίζουμε ιδιαίτερα στο αντικείμενο των οδικών μεταφορών. Βεβαίω είναι και πολύ μεγάλο το δυναμικό και τη εσωτερική ναυσιπλοεία. Στην περαιτέρω διαδικασία επεξεργασία τη έκθεση θα συμπληρώσω με θέματα εσωτερική ναυσιπλοεία. Εν τέλει πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχουν πολλά που πρέπει να δούμε. Η δημιουργία των δικτύων εφοδιασμού πρέπει να είναι σημαντική εναλλακτικά μοντέλα από τους κατασκευαστές, υψηλότερη, φιλο, υψηλότερη φιλοδοξότερη στόχη των χωρών μελών και υποστήριξη των τεχνολογιών αυτών του μέλλοντος από τις χώρες μέλη. Αυτά για την ώρα και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ερτουκ για την παρουσίαση της εκθεσής σας. Πολύ ενδιαφέρουσα και χρήσιμη βέβαια για το μέλλον κυρίως της αυτοκινητοβιομηχανίας και γενικότερα της βιομηχανίας. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σελίνη. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Η προέλευση αυτής της πρωτοβουλίας, όπως θύμισε και ο εισηγητής, είναι η δυσκολία να εφαρμοστεί η οδηγία. Το βασικό πρόβλημα υπογραμμίστηκε και καθορίστηκε από το πώς αντέδρασαν οι χώρες μέλη με διαφοροποιημένο τρόπο. Κάποιες φορές δεν αντέδρασαν καν απέναντι στην ε, ε, έκκληση αυτής της οδηγίας και πιστεύω πως η θέση του εισηγητή είναι σωστή στο, ε, στα όσα λέει αλλά και στη, ε, πώς θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγάλο βαθμό. Συγκεκριμένα νομίζω πως σωστά εντάσσεται στην πρόταση του εισηγητή η ανησυχία την οποία συμμερίζομαι να σεβαστούμε αυστηρά την αρχή της ε, τεχνολογικής ε, ουδετερότητας. Είναι αλήθεια και πρέπει να επαναληφθεί ότι για να ευνοηθεί μια πραγματική διαδικασία ε, μείωσης του άνθρακα θα πρέπει η Ευρώπη και οι χώρες της να έχουν τις υποδομές που διευκολύνουν το ζήτηση από τους καταναλωτές, διότι ο καταναλωτής επιβαρύνεται στην απόφαση αγόρας ε, οχημάτων μικρών ε, εκπομπών, χαμηλών εκπομπών, όταν ξέρει πως δεν υπάρχουν κατάλληλες υποδομές που, που στηρίζουν αυτή του την επένδυση. Από την άλλη πλευρά είναι σωστό να πούμε ότι η διαδικασία απαγόρευσης της του άνθρακα θα πρέπει να ε, παρακολουθείτε με τη λογική και όχι με το να ερωτευτούμε μια μόνη τεχνολογία, μια μόνη τεχνολογική λύση. Οπότε το θέμα αυτό θα πρέπει ε, να το στηρίξουμε. Ε, άλλα στοιχεία επί των οποίων πρέπει να συζητήσουμε, ας πούμε, το οικονομικό θέμα ε, που αναφέρεται με τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ταμείου για την καθαρή κινητικότητα που θα ε, πρικοδοτηθεί με 25 εκατομμύρια μέχρι το 2025. Ε, δεν ξέρω αν θα είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα συγκεκριμένο ταμείο, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι πεπισμένος ότι μέσα στο ΣΕΦ, στη διευκόλυνση για τη ε, ε, Ευρώπη να περιλαμβάνεται και αυτός ο στόχος. Τώρα, όσον αφορά τους στόχους, θα ήθελα να ζητήσω την διαθεσιμότητα του εισηγητή, γιατί όπως συχνά συμβαίνει, ε, ο ορισμός συγκεκριμένων στόχων ενεργοποιεί προστατευτικές αντιδράσεις από πλευρά των χωρών, που συχνά διακόπτουν καν τη συζήτηση και ε, τελικά αυτό έχει αρνητικό αντίκτυπο στον καλό αρχικό στόχο που είναι σε αυτή την περίπτωση η πραγματική εφαρμογή της οδηγίας. Θα είχα να προτείνω λοιπόν μεγάλη προσοχή σε αυτό το, στόχο, σε αυτό το μέσο των υποχρεωτικών στόχων, να μας κάνει να χάσουμε από ε, τον βασικό στόχο, όπως έχει συμβεί παλιότερα. Τώρα, κάτι άλλο που υπογραμμίζει ο εισηγητής όταν αναφέρεται συγκεκριμένα στην στρατηγική που συνδέεται με το πρόγραμμα δράσης για την βιομηχανία των συσσωρευτών μπαταριών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Νομίζω πως είναι σωστή η πρόταση. Το ακούσαμε με τη τρίτη δέσμη για την κινητικότητα στην περασμένη ολομέλεια που, που μας παρουσίασαν ε, Μπούλτς και Κανιέτε, αν θέλουμε να παραμείνουμε πρωταγωνιστές στη διαδικασία της ε, μείωσης της χρήσης του άνθρακα, ε, για, αν και έχουμε μία προσέγγιση μεταβατική, θα πρέπει να έχουμε μια συγκεκριμένη και σοβαρή θέση όσον αφορά το κατασκευαστές συσσωρευτών, γιατί αυτό θα μας επιτρέψει να παραμείνουμε πρωταγωνιστές και, από την υπηρεσία, και για την υπηρεσία και για την παραγωγή και κυρίως θα μας επιτρέψει να δώσουμε νέα διάσταση στο κοινωνικό αντίκτυπο που μπορεί να έχουν αυτές οι μετατροπές στην αγορά εργασίας στην Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή μια δομή της αυτοκινητοβιομηχανίας η οποία θα πρέπει να μας βρει συνεργούς έτσι ώστε στην, στο τέλος της μετάβασης να υπάρχει και μια βιομηχανία του ορεφτόν που θα είναι έτοιμη να δεχτεί όλους τους πολυάριθμους και εξαιρετικούς εργαζόμενους σε αυτόν τον κλάδο. Νομίζω λοιπόν πως τα θέματα που αντιμετωπίζονται είναι σωστά, η γενική προσέγγιση είναι κοινή και γι' αυτό και υπάρχουν έτσι οι προδιαγραφές για εξαιρετική εργασία. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, κύριε Δεσμάκερ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Πρώτα απ' όλα και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εκθεσή του αυτή. όπως λέει και η Επιτροπή, πρέπει πολλές χώρες μέλη να κάνουν παραπάνω προσπάθειες για να περάσουμε σε αυτό τον χώρο κινητικότητας χωρίς άνθρακα. Σωστό. Όμως αυτή η αλλαγή είναι πολύ σημαντική όχι μόνο για να πετύχουμε τους στόχους μας για το περιβάλλον, να τηρήσουμε τη συμφωνία δηλαδή, αλλά για να αντιμετωπίσουμε και, την, ε, και τον παγκόσμιο ανταγωνισμό. Αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να παίζει κάποιο ρόλο στην αυτοκινητοβιομηχανία, τότε θα πρέπει να προχωρήσουμε και να στηρίξουμε αυτά τα αναλλακτικά οχήματα, γιατί μόνο τότε θα μπορέσουμε να τα καταφέρουμε στον ανταγωνισμό μέσω γνώσης, τεχνολογίας κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι πρώτα απ' όλα η κυβερνήσεις μας σε όλα τα επίπεδα πρέπει να προσφέρουν βεβαιότητα, σταθερότητα στον καταναλωτή αλλά και στον κλάδο. Και το έχουμε πει ότι πολλές χώρες μέλη δεν τα έχουν καταφέρει γιατί δεν υπάρχει εθνική πολιτική, δεν υπάρχει ηγετικός ρόλος που είναι πολύ σημαντικός για να μπορεί κανείς να έχει αξιόπιστα προγνωστικά για το μέλλον. Μόνο έτσι μπορούμε να έχουμε και ιδιωτικούς παράγοντες που θα ενισχύσουν αυτήν την αλλαγή. Και δεν πρόκειται μόνο για τη χρηματοδότηση. Και οι εθνικές κυβερνήσεις και οι περιφερειακές μέσω ε, μέτρων μπορούν να καταφέρουν πολλά. Ε, για παράδειγμα, για τις μακροχρόνιες συμβάσεις με διάφορους παράγοντες. Αν υπάρχουν τέτοιες συμβάσεις μακροπρόθεσμες, μπορούμε να προσφέρουμε να συμπεριληφθούν και υποδομές. Υπάρχουν οι χώρες λοιπόν οι οποίες θα ακολουθήσουν αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και αυτό θα αποτελέσει παράδειγμα και για τους υπόλοιπους. Και θέλω να αναφερθώ λιγάκι και στην ενεργειακή ουδετερότητα. Να είμαστε προσγειωμένοι, να είμαστε ρεαλιστές. Η αλλαγή σε μια κινητικότητα χωρίς ε, εκπομπές θα πάρει χρόνο και πρέπει να βρεθούν στο μεταξύ ενδιάμεσες λύσεις αναφέρθηκε στη τεχνολογία υδρογόνου για παράδειγμα, αλλά υπάρχουν και άλλες. Αυτές οι ενδιάμεσες λύσεις πρέπει να εξεταστούν. Προσβλέπω σε επικοδομητική συνεργασία με όλους τους συναδέρφους πάντως. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Ντεμεσμάκερ. Ο κύριος Ρικέ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κι εγώ. Πολύ σύντομα λοιπόν θα μιλήσω εγώ εκ μέρους της Γεζίν η οποία χρειάστηκε να φύγει να πάει σε μια άλλη κοινοβουλευτική επιτροπή, όπου είναι και εκεί η για, ένα, για μια νομοθετική πρόταση. Πάντα είναι πρόβλημα αυτή η επικάλυψη. Λοιπόν, πολύ σύντομα, τι λέει. Λέει ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρεία συμφωνία που και θεματικά και γεωγραφικά να είναι ευρεία και η Επιτροπή θα έπρεπε να δραστηριοποιηθεί ακόμα περισσότερο για το θέμα. Όπως είπε και ο Ισμαήλ πριν, πρόκειται για μια έκθεση πρωτοβουλίας. Έκθεση πρωτοβουλίας που σημαίνει μέτρα επιχειρησιακά από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συνεπώς, χρειάζεται και να επιταχύνουμε και να δράσουμε ουσιαστικά για το θέμα. Τώρα τα κονδύλια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, 800 εκατομμύρια έχει διαθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρξει η ισορροπία με τα δισεκατομμύρια που είχαν προβλεφθεί αρχικά. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεδομένων των όσων προτάθηκαν για τον μελλοντικό προϋπολογισμό, και πιο συγκεκριμένα για τις μεταφορές και το διευκολύνοντα στην Ευρώπη, δεν είμαι πολύ αισιόδοξο για το τι θα πάρουν τελικά οι μεταφορές. Δεν θα υπάρξει μετάβαση εντός εισαγωγικών, ενεργειακή μετάβαση στις οδικές μεταφορές, αν δεν υπάρξει αλλαγή και στο δίκτυο ε, υποδομών και καυσίμων. Αν οι οδηγοί οι χρήστες γενικά δεν είναι εξασφαλισμένοι ότι κάνουν τη σωστή επιλογή αγοράζοντας ένα εναλλακτικό όχημα με εναλλακτικά καύσιμα, δεν θα το κάνουν. Οπότε πρέπει γρήγορα να προχωρήσουμε με αυτή την έκθεση πρωτοβουλίας και να χρησιμοποιήσουμε και τη φαντασία μας όσον αφορά τον προπολογισμό και τα επιχειρησιακά μέτρα. Τέλος η Γεζίν χαίρεται που μπορεί να συνεργαστεί με τον Ισμαήλ για ένα θέμα πάνω στο οποίο, από ό,τι φαίνεται, συμφωνούν επί τη αρχής πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Ρικαίο. Ο κύριος Τέιλορ τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εισηγητή για την έκθεση αυτή. Και εγώ ήμουνα σκιώδη το 2014 εκ μέρους των Πρασίνων για την ε, έκθεση αυτή στην οποία αναφέρθηκε ο εισηγητής που στο τέλος δεν στηρίξαμε. Γιατί διαφωνήσαμε ότι κοινοτικά χρήματα θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν και δημόσιο χρήμα για επιπλέον υποδομές. Πιστεύαμε, όπως και ακόμα πιστεύουμε, ότι δεν μπορείς να υποχρεώσεις τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν αυτοί, αυτές τις υποδομές με επενδύσεις και ότι περισσότερα θα έπρεπε να έρθουν από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτοί πρέπει να προσφέρουν έτσι καλλιώ τις υπηρεσίες, οπότε αυτοί πρέπει να βάλουν και το χέρι στην τσέπη. Χαίρομαι όμως που βλέπω ότι καταλαβαίνουμε πως τα εναλλακτικά καύσιμα δεν σημαίνει ότι από μόνα τους θα βοηθήσουν. Και αυτό ακριβώς το τι θα βοηθήσει την μείωση των εκπομπών στις οδικές μεταφορές είναι αυτό που πρέπει να μας απασχολεί. Χαίρομαι λοιπόν που ο κύριος Σερτούκ αναφέρθηκε στην αυξανόμενη χρήση των εσωτερικών υδάτων και του σιδηρόδρομου, που όντως έχουν πολύ λιγότερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Επίσης γνωρίζουμε ότι ο κύριος Σερτούκ ζητάει μεγαλύτερη στήριξη για τους συσσωρευτές και τις κυψέλες καυσίμων. Όντως είναι μια διέξοδος αλλά πόσο γρήγορα μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Και τι επίπτωση θα έχει αυτό στην ανάπτυξη κυψελών καυσίμων. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Γι' αυτό λοιπόν και για πολλούς άλλους είμαι λόγους, είμαι υπέρ της ενεργειακής ουδετερότητας. Και δεν πρόκειται μόνο επειδή στηρίζω τα ηλεκτρικά ποδήλατα που στις πόλεις αποτελούν ένα εξαιρετικό τρόπο μεταφοράς. Η ηλεκτρική κινητικότητα με εναλλακτικές πηγές ενέργειας βέβαια και όχι με ορυκτά είναι η καλύτερη ιδέα. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Κύριε Κονζάλη, εσεί έχετε τον λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ ε, τον εισηγητή για το έργο του. Είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε πολύ γρήγορα, δηλαδή να μην έχουμε πια άνθρακα στα καύσιμά μας, να έχουμε καθαρά οχήματα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σε μια κατάσταση όπου έχουμε καθυστερήσει φοβερά γιατί από τα όλα τα σημεία, τα 100.000 που είχαμε αποφασίσει για σταθμούς φόρτισης, έχουμε, μάλλον από τα 800.000 έχουμε μόνο 100.000 αυτές τις σημεία φόρτισης. Άρα η κάθε χώρα θα έπρεπε να φροντίσει να τηρήσει την οδηγία του 2014 με σταθμούς φόρτισης και τις εναλλακτικέ πηγές Αλλιώς θα έχουμε κάνει το ίδιο λάθος δύο φορές. Τώρα το έγγραφο που μας παρουσιάζει σήμερα ο κύριο Σερτούκ πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όμως θεωρώ ότι θα μπορούσε να εμπλουτιστεί κατά πολύ. Κυρίως εγώ θέλω να υπογραμμίσω το στόχο του να έχουμε ένα επαρκές δίκτυο σταθμών φόρτισης με καθαρή ενέργεια. Αυτό είναι μια ευκαιρία προκειμένου η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από πολλά χρόνια, από δεκαετίες δηλαδή, να αποκτήσει τη συνήθεια του βιομηχανικού σχεδιασμού. Από πλευρά τη ομάδα μου θα υποβάλουμε τροπολογίε προς ε, αυτό το στόχο του στρατηγικού σχεδιασμού και προκειμένου οι δημόσιε διοικήσει και ο ιδιωτικό τομέα να συνεργαστούν μεταξύ του. Είναι πολύ σημαντικό οι υποδομέ του δημοσίου και του ιδιωτικού να υιοθετήσουν το στόχο αυτό των καθαρών μεταφορών. Υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες εμπορικές εγκαταστάσεις, είτε πρόκειται για ξενοδοχεία, είτε πρόκειται για σταθμούς μεταφορών, στάδια, νοσοκομεία κλπ. κλπ. που θα μπορούσαν να προσαρμοστούν προς αυτή την κατεύθυνση. Έπειτα η στρατηγική τομή θα πρέπει να είναι στην πρώτη γραμμή, να δίνουν το καλό παράδειγμα και έτσι να κινητοποιούνται και οι υπόλοιποι προς τη σωστή κατεύθυνση. Άρα πρέπει να υπάρχει μια σαφής δημόσια πολιτική μεταφορών που να δίνει κίνητρα και στους υπόλοιπους να ακολουθήσουν. Να είναι καθαρές οι δημόσιες μεταφορές και φυσικά να υπάρχουν, ε, όπως είπαμε, σταθμοί επαρκή φόρτισης. Πρέπει να είναι και δεσμευτικοί αυτοί οι κανόνες. Συγχρόνως όμως πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί. Οπότε Ας αρχίσουμε από τα έργα υποδομών στα αστικά κέντρα, όπου υπάρχουν μεγαλύτερα προβλήματα ρήπανσης του αέρα, και να θέσουμε και κάποιες βασικές γραμμές για το πώς θα είναι αυτή η σταθμή φόρτισης. Θα πρέπει να είναι ασφαλής για την υγεία και τις μεταφορές, θα πρέπει να είναι απλή στη χρήση και προσβάσιμη και για τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, θα πρέπει να είναι ανθεκτική αυτή η σταθμή, να μην ε, χαλάνε εύκολα και να είναι και διατροπική και από την άλλη μεριά το έχω πει και άλλη φορά εδώ όλα τα αναλλακτικά καύσιμα δεν είναι ίδια. Δεν είναι το ίδιο να έχουμε φυσικό αέριο από χιλιόμετρα που έχουν χτιστεί με συνεχιζόμενες και επαναλαμβανόμενες παραβιάσεις των, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και άλλα καύσιμα από εναλλακτικέ πηγές ενέργειας που ρηπαίνουν μηδέν. Εννοείται ότι πρέπει να ακολουθήσουμε το δεύτερο δρόμο. Αυτές είναι οι ιδέες μας, λοιπόν, για να προχωρήσουμε με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ, κυρία ο κύριος Κόρ. Κόχ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ ιδίω τον Ισμαήλ Ερτούγκ για τις εξαιρετικές προτάσεις του. Γνωρίζω βέβαια καλά το πρόβλημα του πόσο περιορισμένη είναι η έκταση των εκθέσεων ιδίας πρωτοβουλία και αντιλαμβάνω πολύ καλά το πρόβλημά σου. Με ενδιαφέρει επίση να είμαστε ουδέτεροι σε ό,τι αφορά την τεχνολογία και σε ό,τι αφορά την κίνηση των οχημάτων, αλλά και για τη δυνατότητα να λειτουργήσουν και οι υπόλοιποι τρόποι μεταφορών. Διότι κάθε τρόπο μεταφορών έχει και τα καλά του, έχει και τα κακά του. Ε, με ενδιαφέρει λοιπόν ο πολυμορφικός, ο πολυτροπικό, ε, οι πολυτροπικέ μάλλον μεταφορές. Και σε ό,τι αφορά τώρα τις ε, υποδομές, αυτό βεβαίως έχει σημειώσει μεγάλη καθυστέρηση. Πρέπει να διαπραγματευτούμε λύσει με τι χώρε μέλη, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει από το επίπεδο των Βρυξελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται να αναπτύξουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες δομές επιχειρηματικές. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη στην χρηματοδότηση των υποδομών και να μην τα αφήσουμε όλα στους κατασκευαστές, ούτε να τα απαιτήσουμε όλα, να τα χρηματοδοτήσουν όλα οι κατασκευαστές. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Φώστερ. Ευχαριστώ τον εισηγητή, κυρία Πρόεδρε. Βεβαίω, πολλά ενδιαφέροντα έθεσε στην έκθεσή του. Είχαμε κάνει και μια λεπτομερή συζήτηση το 2014 στην παρούσα Επιτροπή Μεταφορών, όταν είχε έρθει οδηγία. Προφανώς έχουμε χώρες μέλη που δεν τηρούν τις συμφωνίες που έχουν συνυπογράψει. Ποιε είναι άραγε αυτές. Θα ήθελα να το γνωρίζω, διότι θα έχουμε τότε περισσότερη, καλύτερη μάλλον αντίληψη, διότι από το 2014 που έγινε η συμφωνία και έχουμε φτάσει το 2018 δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Αν και δεν συμφωνώ απόλυτα με τον Ερτούκ, όταν εξετάζει κανείς το θέμα, οι χώρες μέλη έχουν και διαφορετικές απαιτήσει. Αντιμετωπίζουν δηλαδή διαφορετικές απαιτήσει. Και για παράδειγμα, ε, η προμήθεια των καυσίμων είναι διαφορετική για τι διάφορε χώρε μέλη. Και γι' αυτό είχαμε αφήσει τι χώρε μέλη να καθορίσουν ε, τι τι ε, ενδιαφέρει και τι τι συμφέρει. Γνωρίζουμε βεβαίω ότι η πιο πολλή ρήπανση συμβαίνει στα αστικά κέντρα. Συχνά όμως δεν λαμβάνουν υπόψη καν και τι μεγάλε περιοχέ τη υπαίθρου, όπου στην πράξη δεν θα μπορεί να σταματά ο καθένας ανά παν χιλιόμετρο, σε κάθε χιλιόμετρο για να ε, φορτίζει το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο. Εν πάση περιπτώσει, οι χώρες μέλη είναι αυτές οι οποίες σε τελική ανάλυση θα πρέπει να αποφασίσουν πώς θα διαμορφώσουν την υποδομή ανεφοδιασμού και ως θα πληρώσει για αυτήν. Θα πληρώσει ο φορολογούμενος μέσω της γενικής φορολογίας. Δεν μπορώ να φανταστώ η, η Επιτροπή Υπολογισμών συγγνώμη, προϋπολογισμών να διαθέσει μερικά δισεκατομμύρια ακόμα για ε, τη δημιουργία υποδομών ανεφοδιασμού. Όπως, είπατε, όπως είπα πριν, άλλωστε το ζήτημα της υπαίθρου είναι το πιο σημαντικό. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι one size fits all. Πάλι, πάντα μπορεί να έχει κανείς υψηλότερους και φιλοδοξότερους στόχους. Αν θέλουμε απαραγμένη από καυσαέρια άνθρακος, το καλύτερο τότε είναι η πυρηνική ενέργεια. Έχουμε όμως χωρίς μέλη που δεν έχουν εν, πυρηνική ενέργεια, πυρηνικά εργοστάσια. Βεβαίω έχουμε και άλλε που έχουν. Η Γαλλία για παράδειγμα. Και μάλιστα, ε, Madame la Présidente, και στο Λονδίνο αγοράζουμε ηλεκτρική ενέργεια από την ΕΔΕΦ τη γαλλική, ε, τον γαλλικό οργανισμό ε, παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματο από πυρηνική ενέργεια. Τέλο πάντων, από κάπου θα πρέπει να προέλθει η ενέργεια αυτή, ακόμα και η ηλεκτρική ενέργεια που θα φορτίζεται ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Βεβαίω να αναζητήσουμε εναλλακτικέ επιλογές. Εγώ δεν υποστηρίζω καθόλου την ιδέα food for fuel, δηλαδή ε, ε, καύσιμα από γεωργικά προϊόντα. Αυτό που θα πρέπει ωστόσο είναι να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Η έρευνα που αρχίζει τώρα για εναλλακτικά καύσιμα για όλους τους τρόπους μεταφορών, βεβαίως και είναι κάτι το οποίο είναι ε, σημαντικό και πολύ ενδιαφέρον. Ωστόσο να είμαστε πιο αισιόδοξοι και πάντοτε να μην χάνουμε, ποτέ να μην χάνουμε τους στόχους μας από τα μάτια μας. Πάντως ευχαριστώ και πάλι τον κύριο Τούκ για την προσπάθεια που έχει καταβάλει. Σας ευχαριστώ κυρία, ε, κυρία Φώστερ, με Κυρία Φώστερ, σας πληροφορώ ότι όντως η Γαλλία είναι χώρα πολύ πυρηνικοποιημένη. Όμως το καλό νέο είναι ότι η γαλλική εθνοσυλλεύση απεφάσισε να μειωθεί το ποσοστό τη ατομική ενέργεια. Άρα και εμεί αναζητούμε εναλλακτικές επιλογές για την ενέργεια αυτή. Μόνο το είπα αυτό προ ενημέρωσή σα. Η ε, κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ορίστε κυρία Αγιάλα Σέντερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον ε, εισηγητή Ερτούγ για αυτή την εξαιρετική πρωτοβουλία που σήμερα, τη στιγμή που πρέπει να συζητήσουμε τον επόμενο προπολογισμό και το στο δημοσιονομικό πλαίσιο, επιβάλλει μια ανάγκη επιταχυντή, δίνει μια χαρακτήρα κατεπήγοντα. Γιατί βλέπουμε πως και η ε, βιομηχανία επιταχύ, πρέπει να επιταχύνει και, οι συσσωρευτές και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αυτά που λειτουργούν με υδρογόνο λειτουργούν ήδη εδώ και χρόνια. Και ε, για να υπάρχει αυτή η αλλαγή και ξέρουμε πως υπάρχει η δυνατότητα να αλλάξει η βιομηχανία μας με μαζικό ε, τρόπο. Γι' αυτό και πιστεύω πως η πρόταση του κυρίου Ερτούγ είναι ε, πολύ χρήσιμη και κέρια και επίκαιρη και απαραίτητα. Εγώ θα ήθελα να θέσω κάποια στοιχεία τα οποία σίγουρα θα είναι σημαντικά. Πρώτον, ε, ανάγκη να διατηρηθεί η πολυμορφία δηλαδή, ε, γιατί έχουμε μεγάλες ε, πόλεις ή ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, ζώνες όπου χρειάζεται να υπάρχει δυνατότητα κανείς να φορτώσει την μπαταρία του ακόμα και στο σπίτι του. Υπάρχουν ε, όμως περιπτώσεις όπου αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό και υπάρχει ε, φόβος, ε, επικρατεί κάποιος φόβος. Ε, μεταξύ των δημάρχων να τοποθετήσουν ε, σημεία φόρτισης. Χρειάζεται λοιπόν μια κατάσταση όπου να λάβουμε υπόψη την πολυμορφία ε, των πόλων. Επίσης χρειάζονται κοινωνικές προετοιμασίες για να χρειάζεται να ενημερωθούν, να υπάρξει κατάρτιση. Ηλεκτρολόγοι, ναι, οι οποίοι τελειώνουν την κατάρτισή τους για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις ανάγκες και μάλιστα να το κάνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα ώστε να δούμε ποιε θα είναι και οι μελλοντικέ μας ε, δεσμεύσεις. Να έχουμε δηλαδή μια προθεσμία γιατί υπάρχει κόσμος που χάνει τη δουλειά του και που πρέπει όμως εντωμεταξύ να μπορέσει να βρει νέου είδους απασχόληση. Να δούμε λοιπόν πώς μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα μπορέσουμε να κάνουμε τέτοια προσπάθεια μέσα στο πλαίσιο του Connecting Europe Facility, όπως είναι αυτή τη στιγμή ή να δούμε αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και νομίζω πως αυτό μπορεί να είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε και να διευκολύνουμε την αύξηση ε, της χρήσης και το πλαίσιο της χρηματοδότησης της καινοτομία θα μπορέσει να μας βοηθήσει ώστε να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες ε, ήδη έχουν ξεκινήσει βέβαια αλλά να υπάρξουν λύσεις ώστε αυτά όλα σε καινοτομίες να μεταφερθούν σε βιομηχανικό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αγιάλα Σέντερ. Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Ερτούγκ, λέει ο κύριος Μίλτεμπουργκ. Δύο πράγματα θέλω να πω. Το ένα είναι ελευθερία και το άλλο είναι φιλοδοξία. Και δεν νομίζω ότι αυτά τα δύο πάνε απαραίτητα χέρι-χέρι. Φιλοδοξία διότι οι χώρες μέλη, η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ευρώπη πράγματι πρέπει να δουλέψουμε με πολύ περισσότερη φιλοδοξία για να καταφέρουμε να έχουμε κάψιμα με εναλλακτικέ πηγές ενέργειας, ακόμα και αεροπλάνα κάποια στιγμή. Και χρειαζόμαστε εννοείται την κατάλληλη υποδομή γι' αυτό. Να μην καταλήξουμε σε μια κατάσταση έκανε η κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Άρα λοιπόν Αυτά πρέπει να τα λέει η έκθεση. Και έπειτα βέβαια πρέπει να τηρήσουμε και τις συμφωνίες των Παρισίων. Και είναι πολύ ωραία όταν έχει κανείς φιλοδοξία. Αλλά από την άλλη μεριά η θελοντική βάση σε άλλη χώρα μπορεί να επιτευχθεί με κίνητρα φορολογικά για παράδειγμα για να μπορέσουν να υπάρξουν περισσότερα οχήματα με εναλλακτικέ πηγέ ενέργεια. Σε άλλη χώρα μπορεί να μην υπάρξουν τέτοια κίνητρα. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι και ο εισηγητή πρέπει να τα σκεφτεί όλα αυτά. Πώς ε, δηλαδή θα προχωρήσουμε σε νομοθέτηση και χρειαζόμαστε βέβαια και την γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής ΣΥΝΤΑ, έτσι, εσωτερικής αγοράς. Είμαι και εγώ εκεί εισηγητής και συζητάμε για το θέμα της κινητικότητας και των αναλλακτικών πηγών ενέργειας ε, στα καύσιμα. Η Επιτροπή θα πρέπει πριν τα τέλη της χρονιάς να έρθει και να μας πει χρειάζεται νομοθεσία τελικά για να αποφύγουμε τα προβλήματα που έχουμε δει σε άλλους τομείς όπως το roaming. Τέλος, Πρόεδρε. Χρηματοδότηση. Είμαι πολύ περίεργη με την νέα αυτή πρόταση ΣΕΦ, τη Διευκόλυνση για την Ευρώπη. Πώς ε, το βλέπει, πιστεύει ότι η Επιτροπή δίνει αρκετέ δυνατότητες για χρηματοδότηση. Εγώ δεν είμαι σίγουρος. Ίσως χρειάζονται περισσότερα κίνητρα. Πάντως είμαι πάρα πολύ περίεργη μετά την ε, παρουσίαση πώς το βλέπει ο εισηγητής. Και τέλος, στην Ολλανδία διάβασα άρθρα για οχήματα που λειτουργούν με υδρογόνο. Για παν, ε, Ιαπωνέζικης μάρκας, στο Ιώτα. Είναι ένα πολύ βασικό το στοιχείο του ανταγωνισμού στο θέμα αυτό. Οι Ιάπωνε προχωρούν. Εμεί θέλουμε μέλλον για τη δικιά μας αυτοκινητοβιομηχανία. Εάν ναι, τότε πρέπει πραγματικά και στην Ευρώπη να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αλλιώς άλλες ήπειροι θα πάρουν το πρώτο χέρι. Γι' αυτό έλεγα ότι χρειάζεται φιλοδοξία και εφόσον έχουμε φιλοδοξία ίσως υπάρχει λιγότερος χώρος για εθελοντική βάση. Ευχαριστούμε κύριε Φανομίτελμπουργκ. Και στείλτε μας αυτό το άρθρο, εμεί δεν το έχουμε διαβάσει, τουλάχιστον εγώ δεν το έχω διαβάσει, οπότε αν μπορείτε να μα το στείλετε παρακαλώ, το άρθρο σας αυτό. Ο κύριος Ρικέ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Ισμαήλ για την έκθεση του. μη παρατήρηση έχω. Τεχνική φύσεω. Αν δείτε την πρόοδο την ανάπτυξη της χρήσης εναλλακτικών πηγών για τις οδικές μεταφορές, επίγειες μεταφορές, χερσές, πρέπει να προσέξουμε το εξής. Πρώτο παράδειγμα. Η αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων με συσσωρευτή. Ξερχίσαμε, ξεκινήσαμε με πολύ μικρή αυτονομία. Με 100-120 χιλιόμετρα τώρα έχουμε φτάσει σε αυτονομία 300 χιλιόμετρα περίπου. Και πολύ σύντομα θα φτάσουμε στα 600 και 700 χιλιόμετρα αυτονομία. Αυτό βέβαια αλλάζει εντελώ τις απαιτήσει του ανεφοδιασμού. Λέγαμε στην αρχή ότι πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί σταθμοί φόρτισης στους δρόμους, γιατί κάθε τόσο θα έπρεπε να φορτίζονται οι συσσωρευτές. Όταν όμως τελικά η αυτονομία αυξηθεί, τότε η ίδια η φύση αλλάζει. Γιατί δεν θα χρειαζόμαστε τόσο πολλούς σταθμούς φόρτισης με το κόστος που γνωρίζουμε, αλλά καλά θα κάνουμε να πάμε σε ηλεκτρική φόρτιση ε, ταχεία. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Γιατί αν αρχίζουμε με την ηλεκτρική φόρτιση, λαμβάνοντα υπόψη πώς έχουν τα πράγματα σήμερα, κινδυνεύουμε να ζούμε με ψευδεστήσεις, να ξοδέψουμε δηλαδή πάρα πολλά χρήματα για πολλούς σταθμούς φόρτισης στους δρόμους και αυτό δεν θα είναι ούτε αυτό που θα χρειαζόμαστε, ούτε θα είναι αποτελεσματικό. Δεύτερον, Θέλω να πω στη Ματιέ ότι αν πραγματικά το υδρογόνο αναπτυχθεί σύντομα, τότε χρειάζεται και η κατάλληλη υποδομή, η κατάλληλη δηλαδή σταθμή φόρτισης. Πολύ περισσότερο από ό,τι έχουμε προβλέψει σήμερα. Αν λοιπόν υπάρξει πρόοδος και όντως το υδρογόνο θα κοστίζει λιγότερο, θα είναι πιο προσιτό και η αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων συσσωρευτών είναι διαφορετική από αυτή που έχουμε σήμερα. Προσοχή, τι θα προβλέψουμε. Μην προβλέψουμε πράγματα βάσει της σημερινής κατάστασης, γιατί κινδυνεύει να έχει ξεπεραστεί πολύ γρήγορα. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στην έκθεση. Ότι δηλαδή δεδομένων των κονδυλίων, δεδομένου του χρόνου που χρειάζεται για την ανάπτυξη δικτύων. Καλά θα κάνουμε να σκεφτούμε προβλέποντας τι θα συμβεί στο μέλλον. Και να μην κάνουμε με τα σημερινά μόνο δεδομένα, να μην κρίνουμε μόνο με τα σημερινά δεδομένα. Τέλος θέλω να πω στην Επιτροπή ότι με απογοήτευσε η παρουσίασή τη για την διαδεσιμότητα, για τη Ευρώπη και επί τη ουσία αλλά και όσον αφορά του τύπους. Νομίζω ότι η Ευρώπη πρέπει να υποστηρίξει πιο συνεπεί στόχου με περισσότερη συνοχή. Ευχαριστούμε κύριε Ρικέ. Είχα γραφτεί και εγώ στον κατάλογο μιλητών, οπότε παίρνω εγώ τον λόγο. Για να πω στον Ισμαήλ Δερτούκ ότι η έκθεσή του έχει τεράστια σημασία. Κυρίως τη σημερινή εποχή που ασχολούμαστε με το μέλλον διαφόρων ε, βιομηχανικών κλάδων. Και προσοχή, γιατί όταν μιλάμε για εναλλακτικά καύσιμα, εννοούμε τα πάντα και τίποτα. Σήμερα αρκεί να βάλει κανείς τον όρο βιολογικό για να νομίζουμε ότι είναι και κάτι φιλικό προς το περιβάλλον, καθαρό. Όχι, τα βιοκαύσιμα για παράδειγμα, όταν κοιτάξουμε την πρόλευσή τους, διαπιστώνουμε ότι μόνο στη λέξη υπάρχει το βιολογικό. Υπάρχει το φινικέλαιο που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το έχει απαγορεύσει από το 2021. Θα δούμε τώρα κατά πόσο θα συμμορφωθούν οι χώρες μέλη. Γιατί είναι πολύ βλαβερό και για το κλίμα, αλλά και για τις γεωργικές γέες, οι οποίες δεν υπάρχουν για να τροφοδοτούν τα οχήματα, αλλά να δίνουν τροφή στον κόσμο. Τώρα, τα είπε και η κυρία Γιάλα Σέντερ. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κυρία Γιάλα Σέντερ, που δεν πρέπει να ξεχνάμε. Είπατε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορές στις ανάγκες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως για τη συνοχή των ε, περιοχών μας. Δεν έχουν τις ίδιες ανάγκες κινητικότητας η ύπεθρος και η άρα πρέπει να υπάρξει και διαφορετική προσφορά. Πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, κυρία Γιάλα Σέντερ. Το τρίτο που επήγει είναι το θέμα της μετάβασης, της αλλαγής σε ένα νέο ενεργειακό μείγμα που πρέπει να λάβει υπόψη τα 13 εκατομμύρια εργαζόμενων στην αυτοκινητοβιομηχανία. 13 εκατομμύρια μισθωτοί είναι κάτι τεράστιο. Αν δούμε την έκθεση Ερτούκ, αλλά και την έκθεση του κύριου Λυρή, βλέπουμε ότι από τη μια έχουμε την τεχνολογία που προχωρά με τεχνολογία ε, της συνδεσιμότητας, αυτονομία κτλ. Και από την άλλη μεριά έχουμε το ενεργειακό μείγμα. Τέλος. Ναι, πρέπει να βρούμε ένα νέο ενεργειακό μείγμα. Υπάρχουν χώρες μέλη που ήδη δουλεύουν με το υδρογόνο. Η Γαλλία, για παράδειγμα, παρουσίασε ένα σχέδιο έρευνας και καινοτομίας για το υδρογόνο. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη στο ενεργειακό μείγμα όταν μιλάμε για τα ηλεκτρικά οχήματα. Γιατί, γιατί όλοι θέλουμε να βγούμε από τα ορυκτά καύσιμα. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι είμαστε πάνω σε ένα ηφαίστειο όσον αφορά το κλίμα. Δεν μπορούμε λοιπόν να θέλουμε να ακολουθήσουμε τους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και από την άλλη να μην κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Η πρόκληση είναι μεγάλη και η φωνή του Κοινοβουλίου παίζει σημαντικό ρόλο για να μπορέσουν να προχωρήσουν και οι χώρες μέλη. Γιατί κολλησιεργούν λίγο σε σχέση με τους προσανατολισμούς του 2014, τώρα έχουμε φτάσει στο 2018, οπότε ελπίζουμε να επιταχύνουν το βηματισμό στο μέλλον. Αυτά από την Πρόεδρο. Κύριε Ντεπρέ, καλώς ήρθατε. Έχετε το λόγο. Καλημέρα σε όλους και σας ευχαριστώ και πάλι για την πολύ πλούσια συζήτηση που έγινε σήμερα. Πολλά σημεία ε, και εισήχθησαν και θα προσπαθήσω να μην σε όλα, αλλά να σας δώσω την προοπτική της Κομισιόν. Καταρχάς και θα ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι Προσπαθούμε να είμαστε αισιόδοξοι καταρχάς. Πιστεύω πως εάν θέλουμε να δείξουμε μια τελείως καταστροφική εικόνα, αυτό δεν θα αντικατοπτρίζει την κατάσταση. Αυτό είναι η πρώτη παρατήρηση. Και επίσης το θέλω να το πω αυτό γιατί σε κάποιες γεωγραφικές περιοχές έχουμε περισσότερους σταθμούς από ό,τι αυτοκίνητα, οχήματα. Είναι μόνο θέμα της πρόσβασης στις υποδομές η απάντηση είναι όχι. Και αν επανέλθουμε στα όσα είπε ο κύριος Ρικέ, συμφωνώ απόλυτα ότι θα ήταν ανόητο να κάνουμε ένα πρόγραμμα με πολύ λεπτομερείς ε, απαιτήσει. να δούμε ποια είναι τα θέματα της πιο πρόσφατης ε, μπαταρίας, του πιο πρόσφατου συσσωρευτή. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε μια πιο συνολική εικόνα, πιο διευρυμένη εικόνα. Αυτό που σίγουρα χρειαζόμαστε είναι περισσότερα οχήματα, κατηγορίες οχημάτων και πιο προσιτά οχήματα. Και τώρα, για να επανέλθω στο όσα είπε ο κύριος Ροκέ... Ε, χρειάζεται να δούμε τι υπάρχει και έχετε δίκιο, ήδη και το αναγνώρισε αυτό όταν είχαμε την προηγούμενη ανταλλαγή απόψεων, ότι να θυμίσω δηλαδή ότι μέσω του προγράμματος στήριξης, μέσω του Connect Europe Facility, στις επόμενες εβδομάδες ελπίζουμε με τα κράτη-μέλη να φτιάξουμε, αλλά και τα κράτη-μέλη θέλουμε να συνεργαστούν μαζί μας, ώστε να έχουμε μια καλύτερη κατανόηση του τι ακριβώς ε, συμβαίνει. Ε, μέσα σε αυτή την έννοια έχουμε πολύ περισσότερα που εμπίπτουν στο εντολή του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής. Και αυτή είναι απάντηση και στην παρατήρηση της κυρίας Γκονζάλος που περνέ, ναι, αλλά πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη νοσοκομεία ε, κέντρα α, καταστημάτων κτλ. Έπειτα, θα έχουμε να κερδίσουμε μόνο από την Ένωση και να επανέλθω του κύριου, στο, στα όσα είπε ο κύριος Εγώ μπορώ να κάνω πρόταση μέχρι το τέλος του χρόνου για την διαλειτουργικότητα των διαφόρων μέσων. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω γιατί οι συνάδελφοι εδώ δίπλα θα με δίνουν. Είναι προτεραιότητα για μας, όχι. Αυτή τη στιγμή δουλεύουμε ε, στο θέμα με διάφορους φορείς. Προσπαθούμε να ξεκινήσουμε δημόσια διαβούλευση όχι με την ιδέα να αρχίσουμε τώρα να προετοιμάζουμε μία συγκεκριμένη νομοθετική διαδήλωση, ε, δήλωση μάλλον, αλλά τουλάχιστον να καταγράψουμε ποια μπορεί να είναι τα εμπόδια, τα προσκόμματα. Τώρα, να επανέλθω σε ένα συγκεκριμένο σημείο ε, και να πω ότι ε, τονίσατε κύριε Ρτούκου το θέμα της ουδετερότητας. Φυσικά δεν έχουμε διαφορετική γραμμή, όχι. Έχουμε την ίδια. Αναφερθήκατε επίσης στη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα ειδικό ταμείο. Εγώ δεν θέλω αυτό να πω παρά το γεγονός ότι βρίσκω ενδιαφέρον πίσω από αυτή την ιδέα είναι ότι είναι ένας τρόπος που ο κύριος Έρτγουτ θέλει να προσπαθήσει να εξασφαλίσει έτσι μεγαλύτερη ε, ασφάλεια και βεβαιότητα και για τους κατασκευαστές, αν δεν κάνω λάθος. Τι κάνουμε λοιπόν από την προοπτική της διευκόλυνσης συνδέοντας την Ευρώπη. Μέσα στο πλαίσιο του νέου PDP σίγουρα θα συνεχίσουμε με τη, τα κονδύλια εκεί όπου χρειάζεται οπωσδήποτε, αλλά βεβαίως θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανάπτυξη εναλλακτικών λύσεων μέσω της διαδικασίας συνδυασμού. Αναφερθήκατε για το, στον προπολογισμό που, θέσαμε στη διάθεση του σχεδίου εναλλακτικών λύσεων, αλλά αυτό δεν αρκεί σίγουρα. Επίσης θέλουμε να υπάρχουν, ε, να υπάρχουν τα κονδύλια και το ίδιο ο, το, κλάδος να μπορέσει να συντονιστεί καλύτερα. Προσπαθούμε λοιπόν να διερευνήσουμε δυνατότητες για τη στήριξη καθαρότερων λύσεων στον τομέα της κινητικότητας. Βεβαίως το ΕΦΣΙ και το InvestEU θα συνεχίσουν να στηρίζουν και να δίνουν όθηση στην κοινοτομία στον τομέα των μεταφορών. Να εξασφαλίσουμε λοιπόν ότι θα υπάρχει συνδυασμός των διαφόρων κονδυλίων και ευκαιριών που θα στηρίξουν τις φιλοδοξίες μας σε αυτό το τομέα. Και να κλείσω με ένα άλλο σημαντικό σημείο που είναι το τι κάνει η Κομισιόν με αυτό το πρόγραμμα. Γιατί δεν έχει προβεί σε πρόταση αναθεώρησης της οδηγίας. Νομίζω πως ήδη σας είπα ποια ήταν η λογική στην προηγούμενη μου παρέμβαση. Να πω λοιπόν ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να μας δώσουν ένα νέο σχέδιο ήδη ε, του χρόνου. Οπότε αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι δουλεύουμε και συνεργαζόμαστε στενά για να προχωρήσουμε σε κάτι πιο αποτελεσματικό για το επόμενό μας ραντεβού. Εάν αυτό δεν αρκέσει, τότε ο συνομοθέτης εν τη σοφία του θα ζητήσει από την Κομισιόν να προβληματιστεί για τις εναλλακτικέ ε, ε, λύσεις. Και θα το κάνουμε δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης. Πιστεύω ότι αν θέλουμε να έχουμε αυτό το επίπεδο φιλοδοξίας και να έχουμε πιο βιώσιμη κινητικότητα θα πρέπει να δούμε τις θέσεις απασχόλησης και την κατάρτιση και αυτό είναι προτεραιότητα για την Επιτροπή μας και γι' αυτό και με χαρά θα συνεργαστούμε μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντεπρέ. Τελευταίο λόγο έχει ο κύριος Ερτούγκο, εισηγητής μας. Πρώτα, ευχαριστώ όλες και όλους τους συναδέλφους και ιδίω βέβαια τους ε, σκιώδης ηγητέ για τι πολλέ ενδιαφέρουσες προτάσεις που περιλαμβάνει στι παρεμβάσει τους. Από τη δική μου πλευρά μπορώ να πω το εξή. Είμαι πολύ ανοιχτός και όσοι με γνωρίζουν, το γνωρίζουν άλλωστε αυτό, άλλωστε πάντοτε, πάντοτε έτσι έπραξα όταν έφερα την ευθύνη μια εκθέσεως και με την ίδια συνεργασία θα προχωρήσουμε και τώρα. Θεωρώ ότι ίσως θα πρέπει να τονίσω κάτι που είπε ο κ. Μίλτεμπεργκ σχετικά με την χρηματοδότηση. Όντως, η χρηματοδότηση είναι περιορισμένη. Τα κονδύλια για τη χρηματοδότηση είναι περιορισμένη. Και είναι περιορισμένα. Και μέσα στα πλαίσια του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια όλοι μαζί. Χρήματα τα οποία τελικώ προορίζονται για το μέλλον και θα αποδώσουν ωφέλεια στη βιομηχανία στο μέλλον να τα διοχετεύσουμε προ την κατεύθυνση αυτή. Εάν δεν κάνω λάθο, σε πολλέ συζητήσει τη προηγούμενη εβδομάδα, και μάλιστα με τον Επίτροπο κ. Χάν, διεπίστωσα ότι σε διάφορα ταμεία υπάρχουν κονδύλια τα οποία προβλέπουν μια σχετική διάσταση. Για παράδειγμα, στα διαρθρωτικά ταμεία υπάρχουν δυνατότητες, και εγώ το γνώριζα αυτό, σε ό,τι αφορά την περιφερική κάλυψη, μπορούν δηλαδή να, αρθούν από εκεί, να αντληθούν από εκεί κονδύλια και να διατεθούν. Το πρόβλημα είναι ότι είναι τόσο κατακαιρματισμένε οι χρηματοδοτήσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ε, ένα εδώ, ένα άλλο εκεί και ούτω καθεξή, ώστε τελικώ γίνεται πάρα πολύ περίπλοκη η υπόθεση αυτή. Η μεγίστη μου παράκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν δεν μπορεί να ξεκινήσει με κατάθεση πρόταση οδηγία, τουλάχιστον να υπολογίσει, να ψάξει να βρει στον προϋπολογισμό ποια επιμέρους τμήματα ε, κονδυλίων ή ταμείων μπορούν ε, να συλλεχθούν ώστε να εξασφαλιστεί πρώτον περισσότερη διαφανεία, δεύτερον λιγότερη γραφειοκρατία και τρίτον να υπάρχει μια ευθεία προσέγγιση. Όταν πρόκειται δηλαδή συγκεκριμένα να πούμε στις βιομηχανίες και εν τέλει στις χώρες μέλη, ιδού υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες χρηματοδότησής σου, να ποια είναι η αρχή στην οποία πρέπει να απευθυνθεί για να εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση, αυτό θα βοηθήσει πολύ. Θα βοηθήσει πολύ να γίνει έτσι. Και εν προκειμένου έχω να απευθύνω την εξή έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κάτι δηλαδή που είδαμε πάλι εδώ στην Επιτροπή Μεταφορών, ότι μεγάλος αριθμός των πολιτικών ομάδων υποστηρίζουν την πορεία αυτή. Μείωση δηλαδή των ε, οξυδίων του άνθρακος με ουδετερότητα τεχνολογική. Με λίγες εξαιρέσεις, αυτή είναι η σύνοψη των απόψεων όσων με υποστηρίζουν. Κάτι που θέλω επίσης να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την παρακαλώ να το λάβει σοβαρά υπόψη, ότι το παρόν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αυτή την άποψη. Μην προσπαθείτε να μας εξηγήσετε ότι εμπιστεύεστε στην δράση των χωρών μελών και θα χρειαστούν άλλα δύο χρόνια μέχρι το 2020, οι οποίες τότε, και σας, αυτή είναι η προφητεία που κάνω, θα μας πούν τότε ότι δυστυχώς οι χώρες μέλη δεν ανέλαβαν τις ευθύνες τους όπως τους ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτά για όσους έχουν χρόνια εδώ ευρωβουλευτές είναι περιττές προσπάθειες. Έχω ξανά και ξανά ζήσει από τις χώρες μέλη να υπονομεύσουν προσπάθειες στραμμένες στο μέλλον και γι' αυτό θεωρώ και λέγω και πάλι εξετάστε Απευθύνομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ποιε χρηματοδοτικέ δυνατότητε υφίστανται ήδη σήμερα, πώ μπορούμε να τι συγκεντρώσουμε. Και δεύτερο, καταθέστε σχέδιο αναθεώρηση ή μάλλον καταθέστε νέα πρόταση οδηγία και μην περιμένετε μέχρι το 2020. Ευχαριστώ και πάλι τα αξιότιμα μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Επιτροπής Μεταφορών. Παρακαλώ, κυρία Σέντερ, δύο λεπτά, ε, δύο δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εκπρόσωπο τη Επιτροπή που πολύ την αγαπάμε. Αλλά είναι η δεύτερη φορά που δεν αισθάνομαι καλά γιατί από αυτά που λέει ε, πραγματικά απογοητεύομαι, είναι αρνητική. Το Κοινοβούλιο είναι υπέρ και πρέπει ακριβώς να χρησιμοποιηθεί αυτή η τάση που υπάρχει ώστε και η Επιτροπή από την πλευρά της να κάνει το δικό της το κομμάτι. Οπότε ελπίζω την τρίτη φορά που θα την ακούσουμε να είναι πιο θετική. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κυρία Γιάλα Σέντερ. Λοιπόν, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 5η 14 Ιουνίου στις 11. Και πριν ε, συνεχίσουμε, θέλω να χαιρετήσω εδώ νέους μαθητές προσκεκλημένους του κύριου Λυρή από το γυμνάσιο 14 με 18 ετών με δύο καθηγητές. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή Μεταφορών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα τους χειροκροτήσουμε, είναι όλοι νέοι, πολύ νέοι και πολύ συμπαθείς. Καλώς ήρθατε. Το μέλλον της νεολαίας είναι στην Επιτροπή Μεταφορών. Συνεχίζουμε λοιπόν και περνάμε στο επόμενο σημείο 8. Παρουσίαση από την Επιτροπή του Εγγράφου Εργασία εκ των υστέρων αξιολόγηση τη επίδοση και των συστημάτων τελών του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Θα μάθουμε λοιπόν για την αξιολόγηση εκ των υστέρων της επίδοσης και των συστημάτων τελών του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. και αξιολόγηση της επίδοσης λοιπόν, αλλά και τα συστήματα τελών, που τα συστήματα αυτά βασίζονται σε δύο εκτελεστικές πράξεις και έγγραφα της Επιτροπής που αποτελούν και το αντικείμενο τη σημερινή μας συνάντηση. Θα δούμε λοιπόν πώς έχει προχωρήσει η εφαρμογή όλων αυτών. Η Επιτροπή θα μας παρουσιάσει το θέμα της και μετά θα πάρουν το λόγο οι ευρωβουλευτές που το επιθυμούν. Στο τέλος θα ξαναδώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή βέβαια για να απαντήσει στα ερωτήσεις και τα σχόλια. Λοιπόν, για να μην καθυστερήσουμε και πολύ, κύριε Καστελέτη, πού είσαστε? Εκεί. Καλώς ήρθατε στην Επιτροπή μας. Έχετε το λόγο για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σε όλους. Όπως είπατε, Πρόκειται για έκθεση της Επιτροπής που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο που μας πέρασε για την εφαρμογή των συστημάτων οτελών του ενίου ευρωπαϊκού ουρανού. Είναι κάτι που αποτελεί μέρος μιας ενιαίας πρωτοβουλίας που άρχισε από το 2000. Πρόκειται για την αξιολόγηση του δεύτερου νομοθετικού πακέτου όσον αφορά τις επιδόσεις για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διάφορες προκλήσεις. Εκαλύπτονται πολλοί τομείς, περιβάλλον, κόστος, αποτελεσματικότητα και το πρόγραμμα αυτό που αξιολογεί τις επιδόσεις είναι βεβαίως να διανεκανοποιούνται αν και τελικοί χρήστες. Το πρόγραμμα αυτό τώρα εφαρμόζεται από το 2011. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε αξιολόγηση των επιπτώσεων του προγράμματος αυτού σε τρία χρόνια. Από το 2012 δηλαδή μέχρι και το 2014. Και μετά υπάρχει και μία δεύτερη περίοδος αξιολόγησης. Κάθε φορά είναι τρία χρόνια. Επόμενη διαφάνεια. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνει πολλές ε, αρχές. Έχει στοιχεία, κριτήρια, έγινε έρευνα που στηρίχτηκε με μια διαδικασία διαβούλευσης. Βλέπετε εδώ τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαβούλευσης που έγινε από εξωτερική επιχείρηση συμμετείχαν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και τελικοί χρήστες και πάροχοι, δίκτυα, συνδικάτα κλπ. Το αποτέλεσμα της μελέτης έδειξε ότι το πρόγραμμα επιδόσεων ανταποκρίνεται στις ανάγκες και αξιολογήθηκε λοιπόν από τους διάφορους εταίρους. Εδώ θα μπορούσα σύντομα να αναφερθώ στο κάθε τομέα επίδοσης. Αποτελεσματικότητα όσον αφορά την ασφάλεια. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι διατηρήθηκαν τα επίπεδα ασφάλειας και μάλιστα βελτιώθηκαν και σε ένα βαθμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπετε εδώ, υπάρχει ο δείκτης ε, επίδοσης στην ασφάλεια. Πόσο αποτελεσματικά λοιπόν είναι τα συστήματα διαχείρισης ασφάλειας. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε τις ικανότητες. Ακόμα και αν ο στόχος αυτός της ικανότητας ε, δεν τηρηθήκε πλήρως, 0,5 λεπτά καθυστέρηση είχαμε αναπτύσσει. Έπεσαν οι καθυστερήσεις όσο γινόταν περισσότερο στην περίοδο 2012-2015 σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Οπότε από τη στιγμή που είχαμε τον νέο ευρωπαϊκό ουρανό μειώθηκαν πολλοί καθυστερήσεις. Και εδώ βλέπετε για την περίοδο 2012-2013. Βλέπετε ότι το 2015 έχουμε αύξηση των καθυστερήσεων. Αυτό έχει να κάνει όμως με την αύξηση και της κυκλοφορίας. Στη συνέχεια για το περιβάλλον. Εδώ υπάρχει ένας δείκτης ο οποίος μετράει το πόσο αποτελεσματικές είναι οι διαδρομές και εδώ βλέπετε ότι υπάρχει βελτίωση. Δηλαδή επέκταξη πτήσεων για λόγους διαχειριστικούς μειώθηκε από το 5.15 στο 4.84. Δηλαδή και εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μια θετική τάση. Όσον αφορά τώρα το τελευταίο τομέα επίδοσης της ε, αποδοτικότητας για το κόστος το κόστος τώρα μετριέται σε πραγματικούς όρους. Και εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπετε ότι το μοναδίο κόστο, το πραγματικό κόστο, μειώθηκε από 59 ευρώ σε, στην κάθε πτήση, το 2015. Οπότε νομίζω και όσον αφορά αυτή τη σχέση κόστους-οφέλους, τα ωφέλη που σας παρουσιάζουμε εδώ δείχνουν και το κόστος του προγράμματος. Αυτό φίλετε όχι μόνο στην απόδοση, αλλά και σε άλλα ρυθμιστικά μέσα, τα οποία χρησιμοποιεί ο ενίος Ευρωπαϊκός Ουρανός, το πρόγραμμα Caesar ή άλλα. Επόμενη διαφάνεια. Εδώ βλέπουμε μία από τις επιπτώσεις εξαιτίας της αύξησης της κυκλοφορίας αποφάσισε η αρχή πάροχων μεταφορών να αναβάλει κάποια δαπάνη επενδύσεις δηλαδή για τον εξυγχρονισμό και η αξιολόγηση δείχνει ότι το πρόγραμμα σωστά αναλαμβάνει το κόστος του συστήματος ελέγχου και τέλος πρέπει να λάβουμε υπόψη μας κάποια στοιχεία που έχουν να κάνουν με την περίοδο αναφοράς που συνεχίζεται, που είναι η δεύτερη περίοδος αναφοράς πρέπει να πούμε ότι οι χρήστες δεν είναι πλήρως ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα γιατί λένε ότι ο συσχετισμός ωφέλους κόστους, τα κέρδη δηλαδή, δεν είναι αρκετά. Όταν υπήρξε ε, τελμάτωση στις μεταφορές δεν είδανε να υπάρχει κάποια βελτίωση. Τώρα αυξάνεται η κυκλοφορία, οπότε πιέζεται το σύστημα πάλι ακόμα περισσότερο. Βλέπουμε ότι αυξάνονται και οι καθυστερήσεις, οπότε θα πρέπει να υπάρξουν επενδύσεις, να υπάρξει πρόσληψη νέων ελεγκτών και περισσότερη ευελιξία όσον αφορά την ικανότητα. Για την επόμενη πεδίο αναφοράς, να ξέρετε ότι εργαζόμαστε για την περίοδο που αρχίζει από το 2020 και θα λάβουμε η υπόψη μας και το τι λέει το ελεγκτικό συνέδριο. Σίγουρα πρέπει να βελτιωθεί η συνέργεια ανάμεσα στο επιχειρησιακό τμήμα και το ρυθμιστικό. Και το πρόγραμμα Caesar και τη διαχείριση. Επίσης, ελέγχουμε και οικονομικές αναλύσεις για να καταλάβουμε καλύτερα τις δαπάνες ανακατηγορία πώς γίνονται αυτές και τι επιπτώσεις έχουν στις επιδόσεις των συστημάτων τελών. Θέλουμε να ενισχύσουμε βέβαια την ελεγκτική αρχή, που τελικά είναι και υπεύθυνη για την εφαρμογή του συστήματος τελών. Και θέλουμε να αναθεωρήσουμε και τους δείκτες. Θα βελτιωθούν και θα χρησιμοποιηθούν νέοι. Τέλος, θα απλοποιήσουμε και το πρόγραμμα για να μειώσουμε το διοικητικό του κόστος. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία λοιπόν και συζητάμε στα διάφορα φόρα, δηλαδή στις χώρες μέλη βάση του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Τελευταία συζητήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και προβλέπεται και άλλη τέτοια συζήτηση τον Ιούνιο. Με στόχο να ολοκληρώσουμε με μια θετική γνωμοδότηση από πλευρά των χωρών ε, μελών το φθινόπωρο. Επίσης θα αρχίσει και συζήτηση για το στόχο όσον αφορά την επόμενη περίοδος αναφοράς από το 2020 και μετά με διαβούλευση με τους διαφορούς ενδιαφερόμενους και απόφαση θα υπάρχει ελπίζουμε πριν τα τέλη της χρονιάς ή πολύ λίγο μετά το νέο έτος για την εφαρμογή του προγράμματος αυτού που κρίνεται επιτυχές. Αυτά και από εκεί πέρα ευχαρίστω να απαντήσω σε ό,τι ερωτήσει έχετε για την πρωτοβουλία αυτή. Ευχαριστώ. beaucoup pour votre intervention et je donne tout de suite la parole à madame. Ευχαριστούμε. Η κυρία Κλούν έχει το λόγο. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον εκπρόσωπο τη Επιτροπή για την παρουσίαση με τα βλέμματα στραμμένα στο μέλλον και σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το σύστημα τελών του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Και βεβαίως η εφαρμογή του πώς υπήρξε. Πάντοτε θέλουμε εμείς να βελτιώνεται η απόδοση των συστημάτων και να συνδέονται τα κίνητρα αυτά και με τα άλλα τμήματα της νομοθεσίας για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό Και αυτό το Joint Undertaking Caesar αναλαμβάνει το ρόλο και ιδίω για τους στόχους αποδοτικότητας. Συμφωνεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ξεχωριστά κίνητρα για την υιοθέτηση του ΣΕΖΑΡ θα πρέπει να μελετηθούν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Γραπίνη. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Παρακολούθησα προσεκτικά τα όσα είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι σαφές ότι χρειαζόμαστε βελτιώσεις. Λέτε ότι κάνατε αξιολόγηση 2012 2012-15 2015 και έχετε παρουσιάσει και ορισμένα δεδομένα. Έχετε συγκεντρώσει δεδομένα από τους operators, από αυτούς που χρησιμοποιούν τον ενέργειο χώρο. Ρωτήσατε τους καταναλωτές. Εγώ πετώ πολύ όλη αυτή τη διάρκεια των ετών αυτών και δεν έχω δει καμιά βελτίωση όσον αφορά την ε, ακριβή άφηξη των αεροσκαφών. Των αεροσκαφών. Έχετε λοιπόν ε, ρωτήσει και τους καταναλωτές, δηλαδή τους χρήστες των υπηρεσιών των αεροπορικών εταιριών. Έχετε κάνει προσπάθεια να αναλύσετε τι προκαλεί τις καθυστερήσεις είτε απλώς σημειώνεται τις καθυστερήσεις στο σύνολό τους. Ως καταναλωτές και καταναλώτριες ενδιαφερόμαστε για την ασφάλεια, για την ακρίβεια, χρονική δηλαδή ακρίβεια των πτήσεων. Είμαι άλλωστε μέλος και της Επιτροπής Προστασίας του Καταναλωτού και με ενδιαφέρει ιδιαίτερω να λάβω κάποιο feedback από εσά για τα ερωτήματα αυτά. Ευχαριστώ κυρία Γκραπίνη, η κυρία Ιούτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή για την παρουσίαση και για την αξιολόγηση που έκαναν μια αξιολόγηση που είναι σημαντική για να δούμε ε, τις προβλέψεις για το μέλλον του ενιαίου ευρωπαϊκού ουρανού. Ε, διαπιστώσαμε το RP1. Δυστυχώς ε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα με προηγούμενη κατάσταση. το ίδιο δεν μπορούμε να πούμε για το RP2 που από ό,τι φαίνεται, μάλλον που δεν μπορούμε να δούμε οριστικά ποιο θα είναι το τέλος. Σίγουρα οι στόχοι και που είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι, υπερβολικά φιλόδοξοι και δεν αντιποκρίνονται στην πραγματικότητα. Πρόκειται μάλλον για πολιτικές αποφάσεις που δυστυχώς δεν βασίζονται σε συγκεκριμένες ε, καταστάσεις που θα μπορούσαν να ισχύσουν ε, ως σημείο αναφοράς για το μέλλον. Θα ήταν ίσως σκόπιμο να έχουμε πιο ρεαλιστική προσέγγιση ε, όσον αφορά την πραγματικότητα και τις οικονομικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτήν. Ε, και πώς ερμηνεύεται στην Κομισιόν αυτό τα αποτελέσματα όσον αφορά την εφαρμογή του επόμενου RP3. Υπάρχουν οι προποθέσει, πληρώνται οι προποθέσει, ή θα έπρεπε να προχωρήσουμε ε, με βάση του σχήματο του δεύτερη, της δεύτερης περίοδου αναφοράς RP2 και σε σχέση με τα αποτελέσματα της δεύτερης αυτής περίοδου που εμπετεύθηκαν ε, και Μόνο μερικά αναφέρουν την αύξηση της κυκλοφορίας. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε μια μεγαλύτερη περίοδο, δύο, τρία, διετή, τριετή, ώστε να λαμβάνουμε υπόψη τα στοιχεία και να τα συγκρίνουμε ανάμεσα στα κράτη. Προφανώς ε, οι στόχοι για τις δυνατότητες, αποτελεσματικότητα, ωφέλεια, κόστος και ασφάλεια, όλα είναι σημαντικά. Όμως βλέπουμε πως δίνεται μεγάλη έμφαση στη μείωση του κόστους, που παρότι είναι απαραίτητο και δίκαιο, δεν ε, θα πρέπει αυτό να έχει αντίκτυπο στην ασφάλεια, για την οποία οι αποταμιεύσεις και οι οικονομίες ποτέ δεν μπορούν να είναι αποδεκτές. Αυτή η σχέση ανάμεσα κόστος και ασφάλεια θα πρέπει μέσα στη τρίτη περίοδο αναφοράς, RP3, να ληφθούν καλύτερη υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γιούτο, κυρία Φώστερ. Ε, τώρα, συγγνώμη, σας ε, δίνω το λόγο τώρα μετά από τους υπόλοιπους. Δεν σας είδα στην αρχή. Εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα, κυρία Πρόεδρε. Δεν, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Και βεβαίως αυτή η εξολόγηση είναι μια ευρωπαϊκή ε, διάσταση σε προοπτική. Δεν μας δίνει όμως πληροφορίες όσον αφορά την απόδοση και πώς θα πάνε μονομενά τα κράτη-μέλη στον τομέα. Όπως γνωρίζετε, ήμουν πρώην εισηγήτρια στη, για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και το υποστήριξα ναι, κάθεν. Όμως, αν αφαιρέσουμε προφανείς λόγους για τους οποίους υπάρχουν καθυστερήσεις, ας πούμε, κακοκαιρία ή διάφορα τέτοια ζητήματα και βέβαια ενδεχομένω υπάρχουν και ε, βλάβες των συστημάτων, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχουμε ωστόσο είναι η ε, συνδικαλιστική ε, αναταραχή. Και ε, αυτό εμπίπτει στι αρμοδιότητε του κράτου μέλου. Μπορεί εμεί να κάνουμε ό,τι θέλουμε, τεχνολογικέ πρόοδου και να σωρό άλλα πράγματα, αλλά δεν είμαστε σε μια θέση όπου βρισκόμαστε, έχουμε κράτη-μέλη Ε, είναι αρμόδια για, άλλα, ε, για τα θέματα τα συνδικαλιστικά και τα εργασιακά. Αυτά επηρεάζουν το κόστος και τον καταναλωτή. Τον καταναλωτή πρέπει να τον αναφέρουμε. Είναι πραγματικά παράδεκτο. Είναι όμως ε, περίπλοκο το θέμα γιατί δεν συμμετέχουμε όλοι μας ε, σε αυτό στις, στις εργασιακές σχέσεις. Αλλά δεν ε, είναι αρκετά καλή η προσπάθεια γιατί δεν βελτιώνονται τα πράγματα. Άρα το δίδαμα που θα έπρεπε από εσά να βγει και να περάσει προς τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν στον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό είναι ότι έχουν και κοινή ευθύνη και ότι δεν πληρούν το δικό τους μέρος όσο θα έπρεπε. Είναι πολιτικά ζητήματα βέβαια και δεν σημαίνει ότι εγώ εδώ που λέω ε, ότι διαφωνώ με το δικαίωμα της απεργίας. Έχω και εγώ συμμετάσχει σε συνδικαλιστικές δράσεις, αλλά πραγματικά αρχίζει να γίνεται γελίο. Και ο αντίκτυπος στον καταναλωτή είναι παράδεκτος. Σα αφήνω λοιπόν να δούμε τι θα πρέπει να κάνουμε. Ξέρω πώ δεν μπορείτε να το σχολιάσετε και τόσο αυτό εσείς από πλευρά της Επιτροπή. Πάντως θα πρέπει να σημειωθεί σοβαρή πρόοδο. Αν δεν γίνει αυτό, ε, τότε θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε τι ευθύνε μα. Ε, εάν θέλουμε να λειτουργήσει ε, θα πρέπει κάτι να, να, να αναλάβουν και τα κράτη-μέλη τι ευθύνε του. Ευχαριστώ, κύριο Βανίντε Μπρόρη, γιατί έχετε εσεί το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ. Μια απλή ερώτηση, γιατί σε ένα από τα κομμάτια της παρουσίασής σας περίοδος αναφοράς είναι 2012 με 2040. Ε, λοιπόν, τι γίνεται με αυτή την ε, περίοδο αναφοράς που είναι η δεύτερη, RP2, πάλι 8 κράτη-μέλη. Και, τι θα κάνετε, ειδικά ε, εκεί που λέει στη δικό σας έγγραφο εργασία ότι οι χρήστες του εναέριου χώρου αναφέρθηκαν στο γεγονός και παραθέτω πως οι στόχοι γενικά δεν ε, υλοποιήθηκαν. Δηλαδή, τα κράτη-μέλη δεν πιέστηκαν αρκετά ώστε να προβούν στι απαραίτητε επενδύσει. Τι θα κάνετε λοιπόν για να του πείσετε να κάνουν τι απαραίτητε επενδύσει, αν. Ε, ε, δεν, ε, δεν βάλουν τις απαραίτητα, τους απαραίτητους πόρους και τις επενδύσεις που πρέπει. Ε, ευχαριστούμε κύριε Βανίτεμπουργκ, κύριε Κόλ. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ ε, την Επιτροπή για την εργασία της. Ε, πιστεύω πως ε, υπάρχει χώρος για βελτίωση γιατί και έχω την εντύπωση από διμερείς ομιλίες και την έλλειψη, υπάρχει, έλλειψη, υπάρχει έλλειψη συνεργασίας ανάμεσα στην ΕΑΖΑ, τον Ευρωκοντρόλ και τις Εθνικές Αρχές Ασφάλειας και θα ήθελα να έχουμε περισσότερη συνεργασία. Ευχαριστώ κύριε Έχω και εγώ μια σύντομη ερώτηση. Στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό είχαμε διαπιστώσει τη δυνατότητα μείωση τη κατανάλωση, κυροζήνης και των ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 10%. Θα ήθελα να ξέρω αν η Κομισιόν έχει πληροφορίες συγκεκριμένες και ενημερωμένες για αυτό το ζήτημα, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενέργεια δηλαδή και το κλίμα. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριε Καστελέτη, έχετε το λόγο ε, για να απαντήσετε ε, και θα είναι περιορισμένος ο χρόνος σας γιατί έχουμε λίγο καθυστερήσει. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομο. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με το, την ανάπτυξη του ΣΕΖΑ, είμαστε μέσα σε αυτό το, τη φάση ε, της έρευνας. έχουμε, ξεκινήσαμε από το 2015 τη φάση ανάπτυξης και βεβαίως αυτό γίνεται και οικονομικά κίνητρα. Συνήθως αυτό, αυτά προέρχονται από το ΣΕΦ, το, την διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Έχουμε δηλαδή εδώ την εφαρμογή λύσεων ΣΕΖΑΡ, που προέρχονται, λύσεις που προέρχονται από την ερευνητική φάση και θέλουμε να εξασφαλίσουμε πως ε, όλες αυτές οι λύσεις αναπτύσσονται με συγχρονισμένο ε, και συντονισμένο τρόπο. Γιατί χρειάζεται συγχρονισμό όταν μιλάμε για έλεγχο ενάρειας ώστε να φτιάξουμε μια νέα επιχειρησιακή έννοια. Δεν μπορεί να είναι διαφορετική κόνσεπτ από το ένα κρατομέλος στο άλλο και εκεί εστιάζονται οι προσπάθειές μας όσον αφορά τα κίνητρα που δίνονται στο project Cesar. Τώρα για τους καταναλωτές. Δεν είχαμε διαβούλευση με τους καταναλωτές. Θα πρέπει να λάβετε υπόψη πως όλα αυτά τα στοιχεία απλά εστιάζουν στην διαχείριση της εναέρειας κυκλοφορίας που είναι υπεύθυνη εν μέρη για κάποιες από τις καθυστερήσεις αλλά ε, το μεγαλύτερο μέρος των καθυστερήσεων οφείλεται στα αεροδρόμια ή στις ε, αεροπορικές εταιρείε και αυτές οι καθυστερήσεις δεν, δεν λαμβάνονται υπαρκώς υπόψη. Φυσικά και υπάρχουν και προβλήματα ε, κακοκαιρία, αλλά είχαμε και πάρα πολλές απεργίες. Ε, αλλά και στη ε, διαχείριση της ενέργεια κυκλοφορίας, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν συμφορήσεις σε κάποια κράτη-μέλη, έλλειψη δυνατοτήτων, γιατί δεν υπάρχουν αρκετοί ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας. που να μπορούν δηλαδή να οργανώσουν την ασφαλή χωρισμό των ε, αεροσκαφών, έλεγχος και ε, χωρισμός του εναέριου χώρου. Αυτό γίνεται από μια ομάδα ελεγκτών και εναέριες κυκλοφορίας. Ε, βεβαίως όλα αυτά θα ελευθούν υπόψη. Υπάρχει το ερώτημα, αυτό το υπάρχον σύστημα το οποίο είναι πολύ δεδρεωμένο, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις επόμενες αυξήσεις της ε, ενέργειας κυκλοφορίας. Δεν είμαστε βέβαιοι ότι το ισχύον σύστημα που βασίζεται σε εθνική βάση ε, θα μπορέσει να ανταποκριθεί στην αύξηση της κυκλοφορίας. Οπότε γίνεται μελέτη για μια νέα αρχιτεκτονική του εναέριου χώρου που θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ελπίζω πριν το τέλος του έτους, ώστε να δείξουμε πως μια διαφορετική οργάνωση του εναέριου χώρου χωρίς σύνορα μπορεί να δώσει περισσότερες δυνατότητες. Φυσικά, η ασφάλεια είναι ε, must, δεν αμφισβητείται η διαχείριση του ενέργειου χώρου παράγει ασφάλεια, παράγει την τον ασφαλή διαχωρισμό και διαίρεση του εναέριου χώρου. Δεν υπάρχει αντίκτυπος σε αυτό το τομέα. Το θέμα είναι κατά πόσο υπάρχει εξάρτηση ανάμεσα στην χωρητικότητα και το κόστος ωφέλες. Δηλαδή πόσο πρέπει να επενδύσουμε στα νέα συστήματα και στους νέους ελεγκτές και κατά πόσο είναι τελογημένο αυτό το κόστος. Θέλουμε να κατανοήσουμε καλύτερα τη σχέση ανάμεσα στην χωρητικότητα και την ε, ωφέλεια σε σχέση με το κόστος όλων αυτών, σε σχέση με την κατάσταση των απεργιών. Ξέρετε πως ε, Γι' αυτά ευθύνονται λίγα κράτη στην Ένωση, αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα. Η Κομισιόν ε, παρουσίασε πέρσι μια ανακοίνωση που έφερε τον τίτλο «Συνδέοντας την αεροπλοεία». Και εκεί είχαμε συνάψει και ένα έγγραφο εργασία της Κομισιόν που εστίαζε την προσοχή στην ε, συνέχιση της διαχείρισης των αέριου χώρου, δηλαδή να υπάρχει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα σε περίπτωση απεργιών, τουλάχιστον να αυληθούν τα, ε, οι επιπτώσεις των απεργιών. Ε, και για να απαντήσω στη ε, στους ε, κυρία Φώστερ και Μπάουζερ, υπάρχουν πολλοί λόγοι. Έλλειψη πολιτικής στήριξης δηλαδή. Χωρίς να υπάρχει στήριξη πολιτικού χαρακτήρα, η πρωτοβουλία ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού δεν θα επιτύχει τους στόχους που θεσπίσαμε πριν 15 χρόνια. Ενδείξεις για την επόμενη περίοδο αναφοράς, RP3, δεν είναι πολλά υποσχόμενες. Η αύξηση της εναέρειας κυκλοφορίας θα αυξηθεί. Ίσως θα έχουμε καθυστερήσεις. Σίγουρα η καλοκαιρινή περίοδος ε, που τώρα ξεκινά τον Ιούνιο θα δούμε τι θα συμβεί, αλλά πάντως αρχικές ενδείξεις είναι ότι οι επιβάτες θα έχουν περισσότερες καθυστερήσεις λόγω της διαχείρισης του αέριου χώρου. Γι' αυτό ίσως θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε την προσπάθειά μας για περισσότερες αδυνατότητες και πιο μεγάλη ευελιξία. Σε σχέση τώρα με τον αντίκτυπο στο περιβάλλον, μιλάμε βέβαια για ένα μικρό τμήμα των εκπομπών, διότι μετράμε τις δυνατότητες παροχής στα αεροσκάφη, τους κανο, λίτερους κανόνες, για να ελαχιστοποιηθεί ε, τις, τις διαδρομές, συγγνώμη, τις ε, συντομότερες ε, διαδρομές και αυτές τις διαδρομές που αφήνουν το μικρότερο αποτύπωμα όμως έχουμε κάποιες δυσκολίες γιατί τα αεροσκάφη τείνουν να πετούν στις πιο βολικές διαδρομές. Δηλαδή πετούν στη διαδρομή που τους επιτρέπει να ελαχιστοποιήσουν το κόστος και για την κυροσύνη και όχι τις ε, διαδρομές που είναι πιο φιλικέ προ το περιβάλλον. Υπάρχουν πολλέ μεταβλητέ που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Να σα ευχαριστήσω για την συμβολή σας και θα δούμε τον επόμενο μήνα τη νέα για την επόμενη περίοδο αναφοράς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καστελέτη. Με λυπεί κάπως γιατί ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος εδώ δεν έχει ληφθεί υπόψη. Ελπίζω λοιπόν προς το μέλλον αυτές οι πτυχές θα λαμβάνονται υπόψη πραγματικά. Ωραία. Έτσι τελείωσε και αυτό το σημείο στην ημερήσια διάταξη. Θα επανέλθουμε έτσι κι αλλιώς σε αυτή τη μελέτη. Ωραία, επόμενο σημείο. Δεν υπάρχουν διάφορα. Οπότε αγαπητοί συνάδελφοι, ραντεβού την επόμενη φορά, Τετάρτη και Πέμπτη, 20 και 21 Ιουνίου. 9 το πρωί, 20 του μηνός λοιπόν. Τελείωσε η συνεδρίαση της Επιτροπής μας περνάμε τώρα σε κεκλεισμένον το θυρόν, Μικρή διακοπή προκειμένου να σταματήσει η μετάδοση στο διαδίκτυο και να βγουν από την αίθουσα όσοι δεν έχουν δικαίωμα να βρίσκονται στην κεκλεισμένον των θηρών συνεδρίαση. Σε 10 λεπτά. Α, σε τρία λεπτά μου λένε. Άντε πέντε. Ωραία. Συμβασμό σε πέντε λεπτά. Μπορείτε να πάτε και για καφέ να φέρετε.